Good Καλώς ορίσατε, συνάδελφοι, μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αρχίζουμε. Μετά την πρωινή μας συνεδρίαση, επαναλαμβάνουμε τις εργασίες μας, όπως βλέπετε, ε, και αρχίζουμε το σημείο 11. Συμπεράσματα της Ουγγρικής Προεδρίας σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και θα ακούσουμε πώς έχει κατάσταση των πραγμάτων στα θέματα ασύλου και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τμήμα των εργασιών της Επιτροπής μας αυτή την εβδομάδα, διότι αφορά τα συμπεράσματα της Προεδρίας, προκειμένου της Ουγγρικής, το Ουγγρικό εξάμεινο, όπου προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουγγαρία, ως γνωστόν, και χαιρόμαστε που έχουμε ενώπιόν μας δύο εξέχοντα μέλη της Ογγρικής Κυβέρνησης. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε. Μεγάλη μας τιμή η παρουσία σας εδώ και προσβλέπουμε λοιπόν να ακούσουμε τα συμπεράσματα της Ουγγρική Προεδρίας τον κύριο Τίμπορντ Ναυράξης που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργό ε, Δημόσια Διοίκηση και δικαιοσύνη πρώτα και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Σάντορ Πίντερ, Υπουργό Εσωτερικών. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ πριν από έξι μήνες, στις 26 Ιανουαρίου 2011 είχα ήδη την ευκαιρία ε, να έρθω στην Επιτροπή σας για να σας μιλήσω για τους στόχους της Ουγγρικής Προεδρίας, τις προγραμματικές δηλώσεις ουσιαστικά. Ε, τώρα ένα εξάμεινο αργότερα βαίνει προς το τέλος της η Ουγγρική Προεδρία και έχω πάλι τη χαρά να βρίσκομαι ενώπιό σας για να σας πω ότι καταφέραμε να φτάσουμε στους σημαντικότερους στόχους που είχαμε θέσει για την Προεδρία μας. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια σύντομα επ' αυτού και στη συνέχεια ε, θα χαιρόμουν πάρα πολύ ε, αν μου κάνατε ερωτήσεις και είχαμε μια συζήτηση επ' αυτό. Όταν ορίσαμε τους στόχους μας λοιπόν για τη δικαιοσύνη, ε, για την Ουγγρική Προεδρία, το σημαντικότερο για μας ήταν ο παράγων άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που θέλαμε ε, ήταν να υπηρετήσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη. Όλοι μας άλλωστε θέλουμε να ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι φιλική προς τον πολίτη και κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη. Για να επιτύχουμε λοιπόν αυτό το στόχο, κάναμε ό,τι μπορούσαμε κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας και τολμώ να ισχυριστώ ότι στέφθηκαν με επιτυχία οι προσπάθειές μας. Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εποχή της θέσεως σε ισχύ της συνθήκης της Αβώνας κατοχυρώνεται πλέον και στο θεμελιώδη χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η συνθήκη ο χάρτης, ενδεχομένως να αποφασίσουμε και περαιτέρω μέτρα. Αρχίσαμε λοιπόν, δρομολογήσαμε ε, τον Ιανουάριο στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το Συμβούλιο μπορούν να προστατεύουν τους Ευρωπαίους πολίτες ε, σύμφωνα πάντα με τη συνθήκη και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το Μάιο ακολούθησαν ε, και επίσημα συμπεράσματα στο Κανονικό Συμβούλιο Πλέον Υπουργών στο τακτικό. Επίσης, το Συμβούλιο τον Ιούνιο ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας στην Ένωση και η δράση της Ένωσης μπορούν να έχουν απτά και χειροπιαστά αποτελέσματα μόνο εφόσον ε, λειτουργούμε πράγματι στοχευμένα και κοντά στο πολίτη για να το ζει στην καθημερινότητά του αυτό ο Ευρωπαίος πολίτης και να το διαπιστώνει ότι η Ένωση κάνει κάτι για αυτόν. Αυτή η κοινοτικοποίηση λοιπόν της ηθαγένειας του Ευρωπαίου πολίτη δεν σημαίνει μόνο ότι τα δικαιώματα αυτά οφείλουν να εφαρμόζονται και ότι μπορεί να προσφεύγουν οι πολίτες στα δικαστήρια, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά επιπλέον δημιουργούμε και μια κοινωνία πολιτών μια κοινότητα πολιτών με την ουσιαστική έννοια και με την έννοια των αρχών και των αξιών, όχι αμυγός τη νομική και την προσφυγή στα δικαστήρια, το τυπικό τη υπόθεση. αλλά έχουμε και μια ουσιαστική ολοκλήρωση. Αυτό το θέμα συζητήθηκε τον Ιανουάριο στο Άτυπο Συμβούλιο με βάση την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ιθαγενή, την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Κάτι άλλο που έχει σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων είναι η ε, ε, πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Συμβασή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην ΕΣΔΑ. Αυτό για μας ήταν προτεραιότητα, έτσι και αλλιώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τα θεσμικά της όργανα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είχαμε και τις τελευταίες ε, τεχνικές συνομιλίες λοιπόν και τώρα βρισκόμαστε σε επίπεδο διαδικασιών ε, νομικών και τυπικών εσωτερικών για να ε, προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλη προτεραιότητα δική μας ήταν η προστασία των θυμάτων αξιόπινων πράξεων. Το Μάρτιο στη Βουδαπέστη διοργανώσαμε και μια διάσκεψη για να δούμε ποια είναι τα βασικότερα προβλήματά τους και να εκπονήσουμε κάποιες προτάσεις για λύσεις αυτό. Μετά τις συζητήσεις λοιπόν που έγιναν σε αυτές τις διασκέψεις, στη συγκεκριμένη διάσκεψη, η Ουγγαρία πρότεινε ένα χρονοδιάγραμμα για την προστασία των θυμάτων που ε, φιλοδοξεί να είναι κατευθυντήρια γραμμή και πάλι και να οδηγήσει ε, σε ένα ποιοτικό σύστημα παροχής, αρρωγής και υποστήριξης στα θύματα εγκληματικών ε, πράξεων. Αυτό το έγγραφο το συγκεκριμένο εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ιστορικών και Δικαιοσύνης και χαρακτηρίζεται ως ατζέντα ή χρονοδιάγραμμα της Βουδαπέστης. Άλλο θέμα, η χρονδιαγραμμα της βουδαπεστης αλλο θεμα η προστασια των δικαιωμάτων των παιδιών. Όσο γίνεται να προστατεύονται τα παιδιά και να μην πέφτουν θύματα εγκληματικών ενεργειών. Και Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, όπως και τα αλλα κρατημέρια, άλλωστε, και η Ουγγαρία δίνει πολύ μεγάλη σημασία και προσοχή σε αυτό το θέμα. Μια απόφαση πλαίσιο κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών και επίσης μια νέα σύγχρονη νομοθεσία Ε, ήταν ε, μέλημα του τρίου της Προεδρίας της ε, Ισπανικής, Βέλγικης και Ουγγρικής. Θα θυμάστε ότι είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια στο Λανσαρότε. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι η συγκίτρια κυρία Αντζελίλη ήταν πάρα πολύ δραστήρια και χάρη σε εκείνη και στους ούγλους συναδέλφους που συνεργάστηκαν πάρα πολύ ε, βρισκόμαστε στα πρόθυρα συμφωνίας και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η νομοθετική διαδικασία θα αρχίσει και μάλιστα όχι μόνο θα αρχίσει αλλά και θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια ακόμα της Ουγγρικής ε, Προεδρίας. Τώρα, η προστασία των μειονοτήτων, η καταπολέμηση της ένδειας και επίσης η βελτίωση, η ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης στο Ρωμά ήταν προτεραιότητες ε, της Ουγγρικής Προεδρίας. Το Μάιο είχαμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στην ανακοίνωση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική για τους Ρωμά και τονίστηκε η πολιτική δέσμευση των κρατών μελών να συμμετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έρχομαι τώρα στην προστασία δεδομένων και θα ήθελα να σας πω το εξή. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα νέο μέσο ενιαίο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με πολλές εκδηλώσεις και διοργανώσεις, επανειλημμένες διαβουλεύσεις, ε, πάντα σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εδώ επιτύχαμε το στόχο μας εγκρίθηκαν συμπεράσματα στο Συμβούλιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ελπίζουμε η διάσκεψη εμπειρογνωμόνων για το θέμα των μελλαντικών προκλήσεων που ε, αρχίζει αύριο να ανοίξει νέους δρόμους. Διαπιστώνουμε ότι οι διαπραγματεύσεις ε, για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν αρχίσει και ε, εμείς τις παρακολουθούμε και τις συνοδεύουμε ε, στο Συμβούλιο σε διάφορες συνεδριάσεις και σε επίπεδα. Έρχομαι τώρα στο ποινικό δίκαιο. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό και το θέμα της ποινική δικονομίας και στη Βελγική Προεδρία και στην Ουγγρική. Η Βελγική Προεδρία είχε δώσει προτεραιότητα στην ενημέρωση των υπόπτων κατά τη διάρκεια των τριμερών ε, διαλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εισηγήτρια την κυρία Σίπελ ε, πετύχαμε σε πολλά σημεία συνένεση αλλά χρειάζεται και άλλη συζήτηση το θέμα αυτό. Θεωρώ σύντομα ότι πρόκειται να συμφωνήσουν το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Χρειάζονται όμως και περαιτέρω διαβουλεύσεις, δεν έχει λήξει. Και επίσης θα ζητηθεί ε, επίδειξη ευελιξίας ε, και ελαστικότητας ε, κατέρωθεν. Νομίζω ότι και το Κοινοβούλιο έχει δείξει προθυμία ε, εξέβρεση συμβασμού και σας παρακαλώ να διατηρήσετε την ίδια στάση και στο μέλλον για να μπορέσουμε να επιτύχουμε. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για μας ήταν ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας. Στις 10 Ιουνίου, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, ε, συμφωνήθηκε καταρχήν η πρόταση και μπορούμε να διαβεβάσουμε στην Πολωνική Προεδρία το φάκελο αυτό προς περαιτέρω συζήτηση για τις ε, ιδιαίτερες διατάξεις, γιατί επί της αρχής έχει συμφωνηθεί. Επίσης, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι κάτι που μας απασχόλησε. Τον Απρίλιο διοργανώσαμε αντίστοιχη διάσκεψη και πρόσφατα στο Συμβούλιο στις 10 Ιουνίου εγκρίθηκε μια κοινή προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά τη δικαστική συνεργασία σε θέματα αστικού δικαίου, ε, θέλαμε να πετύχουμε πρόοδο στον αντίστοιχο κανονισμό, διότι η Υπήρχε μια πρόταση ε, για τις δικαστικές αποφάσεις και για τη διασυνοριακή συνεργασία ε, σε θέματα κληρονομικού δικαίου για τους κληρονόμους και ε, άλλους ενδιαφερόμενους. και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπόδειγμα συνεργασίας και δράσης προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Βελτιώνεται η κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά τα κληρονομικά ζητήματα και αποφεύγονται επικαλύψεις και διπλές διαδικασίες. Ταυτόχρονα όμως έπρεπε να σεβαστούμε ε, την ε, δικαστική και την νομική κυριαρχία του κάθε κράτους. Στο Συμβούλιο Ιστορικών και Δικαιοσύνης επίσης ε, εγκρίθηκε ένα πολιτικό πακέτο συμβιβασμού ας πούμε για το θέμα αυτό. Άλλο θέμα, αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε θέματα εμπορικού ε, δικαίου και αστικού. Ε, η αλλαγή της νομοθεσίας, λεγόμενο πακέτο Βρυξελών 1, ήταν επίσης προτεραιότητα. Ένα σχέδιο κατέθεσε η Προεδρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, ως βάση για τις περαιτέρω εργασίες κωδικοποίησης. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, με χαρά ε, μπορώ να σας δηλώσω ότι κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας σε θέματα δικαιοσύνης καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικές πρόοδους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά για την υποστήριξη και την καλή μας συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ισπανική και τη Βελγική Προεδρία διότι ήταν τα δύο κράτη-μέλη που προετοίμασαν το έδαφος για μας στο τρίο αυτό της Προεδρίας και ε, ήταν πολύ καλό το γεγονός ότι μας διαβίβασαν κάποιους φεκέλες που προχωρήσαμε, προωθήσαμε κι εμείς. Εύχομαι στο επόμενο τρίο Πολωνία, Δανία, Κύπρο κάθε επιτυχία και ε, να είναι βέβαιοι ότι μπορούν να υπολογίζουν στη συνεργασία μας πάντα και στην επικοδομητική στάση της Ουγγαρίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ναυράξης για την παρουσίαση αυτή σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα διότι η προβλεπόμενη εισήγηση και από τους δύο υπουργούς και η συζήτηση προβλέπει, προβλέπεται για μια μισή ώρα, δηλαδή μέχρι τις 4.30. Στη συνέχεια προβλέπεται ψηφοφορία σε σχέση με αρκετές πρωτοβουλίες Γι' αυτό προτείνουμε να ακούσουμε τώρα τον Υπουργό Εσωτερικών, διότι υπάρχουν ε, μέλη που έχουν άλλες υποχρεώσεις και μετά θα αρχίσει η συζήτηση. Ε, καταρχήν θα λάβουν το λόγο οι συντονιστές, ένας από κάθε πολιτική ομάδα και τα υπόλοιπα μέλη σε δύο γύρους ερωταποκρίσεων και απαντήσεων και από τους δύο υπουργούς. Αυτό προβλέπεται μέσα στη μια μισή αυτή ώρα, μέχρι τις 4.30 δηλαδή. Ο Υπουργός, ο κύριος Πίντερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι ενώπιόν σας για άλλη μία φορά για να σας πω λίγα λόγια για το τι είχαμε προετοιμάσει ως Προεδρία και τι επιτύχαμε. Είχαμε ορίσει τους στόχους και τις προτεραιότητές μας, όπως γνωρίζετε, και θα ήθελα να πω ε, εν είδη εισαγωγής ότι τώρα βρισκόμαστε στο τέλος της ε, Προεδρίας, της τριμερούς αυτής Προεδρίας μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και έπρεπε βεβαίως να αρκεστούμε και στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε αρχικά οριστεί και όπως είχαν ορίσει και οι προκάτοχοί μας δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας και συνεργαζόμενοι μαζί σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έπρεπε να προβλέψουμε όλους αυτούς τους ε, παράγοντες Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι ευεργετηθήκαμε αμοιβαία από τη συνεργασία αυτή. Καταρχήν μας απασχόλησε η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Από το 2006, δηλαδή μετά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, κανένας δεν είχε προσδώσει τόσο μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έπρεπε να δούμε τις κοινωνικές αλλαγές που είχαν επέλθει καθώς και τις αλλαγές μεθόδων του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν είχαμε σαφή λοιπόν εικόνα της κατάστασης ούτε τις αλλαγές που είχαν επέλθει από το οργανωμένο έγκλημα και ομάδες. Όμως καταφέραμε να διεκπαιρεώσουμε αυτή την εργασία και έχουμε ένα βιβλίο καθώς και ένα CD τα οποία σας δείχνω τώρα, όπου καθορίζουμε τους στόχους μας και το τι επιτύχαμε. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραν μέρος σε αυτές τις εργασίες, μα μίλησαν για τις εμπειρίες τους με τις αστυνομικές δυνάμεις, εμπειρογνώμονες και ούτω καθεξής. Και έτσι συλλέξαμε αυτά τα στοιχεία και έχουμε αυτό το εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω αυτή τη σειρά αποτελεσμάτων στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό σας τα παραδίδω, ε, Πρόεδρε, πρόκειται για το εγχειρίδιο και το ΣΥΔΙ. Βεβαίω υπάρχουν και άλλα αντίτυπα για όποιον ενδιαφέρεται. Αυτό μας ε, ενδιέφερε ήταν να οικοδομήσουμε αμοιβαία μέτρα εμπιστοσύνης να οικοδομήσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα ήθελα να στραφώ σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Κοέλιος στην έκθεσή του, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στη συνεργασία όταν μιλάμε για έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα και προσβασιμότητα σε αυτά. Αυτό το θέμα ε, τέθη σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο κεκτημένο του Σέγγεν, στο χώρο του Σέγγεν. Φτάσαμε σε αυτά αποτελέσματα και έτσι τα μέλη του Κοινοβουλίου θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Μέσα στα πλαίσια του οργανωμένου εγκλήματος μας ενδιαφέρει και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, χρησιμοποιώντας δηλαδή τις νέες τεχνολογίες. Δέκα χρόνια πριν στη Βουδαπέστη ε, τέθησε εφαρμογή μία συμφωνία, μία σύμβαση η οποία ακριβώς αναφέρεται στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον χώρο. Αρκετές χώρες έχουν μονογράψει τη συμφωνία αυτή. Θα ήθελα όμως να πω ότι υπάρχουν υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία, δεν έχουν μονογράψει τη συμφωνία αυτή. Εδώ προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και η αρχική αυτή συμφωνία ήταν απαράβατος όρος για να φτάσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα πρέπει να επιτελεστεί μεγαλύτερη πρόοδος. Τρεις τομείς ιδιαίτερα μας απασχόλησαν το PNR με τις ε, ε, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία για τα προσωπικά δεδομένα των ε, επιβατών. Με τις δύο χώρες φτάσαμε σε συμφωνία, όχι όμως με τον Καναδά. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τον Καναδά. Επίσης υπάρχουν οι αποφάσεις ε, προυν για τις ε, διασυνοριακές αποφάσεις. Όταν αναλάβαμε την ε, Προεδρία ασχοληθήκαμε με τρία ζητήματα πρωταρχικά. δακτυλικά αποτυπώματα, μητρώα και ούτω καθεξής. Και τώρα βλέπω ότι 15 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει και τις τρεις αυτές συμβάσεις. Στα πλαίσια της απόφασης πριν. και ελπίζουμε και άλλα κράτη να προσχωρήσουν. Θα θέλαμε να ασχοληθούμε με θέματα καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας, διότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου, γιατί πλησιάζει πάλι η, ημερομηνία αυτή. Όπως ξέρετε, είχαμε εξελίξεις με το θέμα ο ΣΑΜΑ και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη ανταλλαγή απόψεων η οποία προχώρησε έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις μετά από την θανάτωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Σε σχέση τώρα με την ε, επέκταση του χώρου ε, Σέγγεν, βλέπουμε ότι γνωρίσαμε πολλές παλινοδίες και γενικά σκαμπανεβάσματα. Θεωρούσαμε ότι αυτό ήταν από τα πρωταρχικά εύκολα καθήκοντά μας, όμως η Βουλγαρία έπρεπε να κάνει ορισμένες προσαρμογές σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές και ακούσαμε από τους Υπουργούς Εσωτερικών της Γαλλίας και της Γερμανίας ότι είχαν μεγάλες ανησυχίες ως προς την προσχώρηση των δύο αυτών κρατών. Μέχρι στις 15 Μαρτίου η Βουλγαρία προσαρμόστηκε ως προς τις τεχνικές αυτές προδιαγραφές και ε, στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης φτάσαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Σεπτέμβριο θα γίνει μια περαιτέρω αναθεώρηση. Οι δύο αυτές χώρες ε, πληρούν τα τεχνικά προαπαιτούμενα και στον τομέα δικαιοσύνης και τις ε, προαπαιτήσεις για τις δύο αυτές χώρες, νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα φτάσουμε στους στόχους μας. Ανήκτυψε και ένα άλλο θέμα σε σχέση με το Σέγγεν. Χρειάζεται μία αναδιάρθρωση έτσι ώστε να έχουμε υψηλότερες προσδοκίες και συμφωνίες. Είμαι πεπισμένος ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των πολιτών ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα ως προς την ε, ε, κυκλοφορία των προσώπων ήταν αυτό και ο χώρος του Σέγγεν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που ελοχεύουν σε σχέση με τα σύνορα Σέγγεν. Πρόκειται για νέες προκλήσεις και ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές. Αυτό ισχύει ε, για εμάς, δηλαδή το αντιμετωπίσαμε και εμείς και θα το αντιμετωπίσει και η Πολωνική Προεδρία. Είδαμε επίσης τι συμβαίνει στην Λιβύη, την Ισία και Αίγυπτο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάστηκε μία τάχιστη και αποτελεσματική λύση με βάση τα πρόσφατα τεκτενόμενα και έπρεπε να συσταθεί ένα κέντρο εποπτείας και πληροφόρησης. Άρα λάβαμε βραχυπρόθεσμα μέτρα και δόθηκε υποστήριξη στα νότια κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στην Ιταλία, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την ε, ευνίδια εισρωή μεταναστών. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το ύψος της υποστήριξης. Άρα υπήρξαν αντιδράσεις και μέτρα και ως προς τη Frontex ήταν τάχιστη η αντίδρασή μας και αυτό το αναγνώρισαν πολλοί μιλήσαμε και για την κατάσταση στη Μάλτα, διότι πρόκειται για μία μικρή χώρα η οποία πρέπει να ανταποκριθεί σε μία πολύ υψηλή πίεση. Γι' αυτό εκινήθηκε ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Και πολλοί πρόσφυγες μετέβησαν σε άλλα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να ε, ε, ελαφρύνουμε κάπως τη Μάλτα. Επίσης, 174 πρόσφυγες επέστρεψαν στο Τσάντ και άλλους 114 τους ανέλαβαν άλλα κράτη-μέλη. Επίσης, προβάλαμε ε, δραστηριότητες και οργανώσαμε πτήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους Ευρωπαίοι πολίτες. Επίσης, θεωρήσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκπροσωπείται σωστά στη Λιβύη. Όπως ξέρετε, η, Ουγγρική αντιπροσωπεία και οι διπλωμάτες παραμένουν in situ. Όταν ε, αρχίσαμε να ασχολούμαστε, να επεξεργαζόμαστε τους στόχους μας, ασχοληθήκαμε και με την Ελλάδα. Ξέρετε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει έκτοτε, διότι και η Κύπρος, Μάλτα και η Ιταλία αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα. Γι' αυτό βρέθηκαν όλες αυτές οι χώρες στην εμπροστοφυλακή. Άρα μας αποσχόλησε το θέμα της χορήγησης ασύλου και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θέτει ως προθεσμία το 2012. Μέχρι τότε πρέπει να έχουμε επιτύχει πολλά. Έχουμε επιτύχει αρκετά αποτελέσματα. Στις 11 Απριλίου στο Συμβούλιο Πουργών εγκρίναμε μια οδηγία σε σχέση με το καθεστώς μόνιμης διαμονής που αποτελεί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Επίσης επήλθε πρόοδος σε σχέση με την οδηγία προδιαγραφών και προσόντων. Επίσης, μετά τη συνδιαλλαγή, ελπίζω την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες σε σχέση με τον κανονισμό του Δουβλίνου έγινε λόγος, όπως ξέρετε, για αναστολή του κανονισμού του Δουβλίνου. Και εξαιτία των γεγονότων στη Βόρεια Αφρική και ιδιαίτερα στη Λιβύη δεν ανεστάλησαν οι διαδικασίες. Ορισμένα κράτη-μέλη ε, χρειάστηκε να δεσμευτούν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα μεταξύ αυτών και, κανένας, ε, δεν έγινε καμία επιστροφή ε, δυνάμει της Συμφωνίας του Δουβλίνου. Και η Ουγγαρία δεσμεύθηκε σε αυτό το τομέα. Ως προς τη Eurodac θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, προσπελασιμότητα στα στοιχεία της αστυνομικής αστυνομικές δυνάμεις και τις ομάδες ε, αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, όσον αφορά την, ε, τις περιπτώσεις επανεγκατάστασης. Το συζήτησα αυτό το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών και προσπαθούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα για τις επανεγκαταστάσεις. Ελπίζω να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Όταν μιλάμε για τον οργανισμό ε, χορήγησης ασύλου, θα ήθελα να πω ότι στις 19 Ιουνίου θα αρχίσει να λειτουργεί αυτός ο οργανισμός και η κυρία Σαρτζεντίνη είχε αποβάλει ε, ένα ερώτημα επί του θέματος. Δεν έχουν ε, ληφθεί αποφάσεις. Θεωρούμε όμως ότι φτάσαμε σε αυτό το πολύ μεγάλο βήμα. Σε σχέση με την ε, νόμιμη μετανάστευση, προσπαθούμε να βρούμε μία και ενιαία παράμετρο αντιμετώπισης του ζητήματος. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Και μέσα στα πλαίσια του άτυπου τριμερούς διαλόγου ελπίζουμε να διασφαλίσουμε τα αποτελέσματα που αποζητούμε σε σχέση με intra-corporate μεταφορές θεωρούμε ότι αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, διότι θα πρέπει οι πολυεθνικές να μπορούν να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην κοινοτική επικράτεια. Δεν μπορέσαμε όμως να φτάσουμε σε τελικά αποτελέσματα. Έχουμε ένα προσχέδιο επιτάπητος και μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση κατάσταση βρίσκεται πολύ κοντά με εκείνη της οδηγίας για τους εποχικούς εργαζόμενους. Σε σχέση με του, τις συντονισμένες εργασίες πολέμηση της παράνομης μετανάστευσης έχουμε εγκρίνει μια στρατηγική και στις, αυτό έγινε στις 9 Ιουνίου και επίσης μας απασχόλησε και ο κανονισμός Frontex. Πρόκειται για ένα θέμα μείζωνος σημασίας που σας απασχόλησε και εσάς. Από όσο γνωρίζω υποβλήθηκαν 300 τροπολογίες και οι 103 υποβλήθηκαν για το Συμβούλιο. Δεν επήλθε λοιπόν συμφωνία, αλλά μπορέσαμε να επιλύσουμε το θέμα ως προς 100. Για τρεις δεν έχουμε διευθετήσει το θέμα. Ελπίζω όμως να το καταφέρουμε στο εγγύς μέλλον για να φτάσουμε σε μία συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Αυτά ήθελα να πω. Εν ολίγης, σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας και τη συνεργασία σας και ελπίζω να θεωρείτε και εσείς ότι η εργασία μας ήταν αρκετά θετική. Αρχίζουμε τις συζητήσεις. Θα ήθελα για να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση εντός του προδιαγραμμένου χρονικού ορίου και επειδή ούτως ή άλλως οι δύο υπουργοί μας έχουν ενημερώσει και γραπτός οπότε έχετε όλοι λάβει τις σχετικές εκθέσεις θα ήθελα να μην ξεπεράσει το δίλεπτο καθένας. Πρώτος γύρος με εκπροσώπους των ε, ομάδων και δεύτερος γύρος πρώτα από το ΕΛΚ ο κύριος Σόγκορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο υπουργούς, Ναυραξίτς και Πίντερ ε, και να τους ευχαριστήσω θερμά για το έργο τους κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Ο κύριος Πίντερ ήδη απάντησε για το Σέγγεν και έδωσε την ημερομηνία του Σεπτεμβρίου, οπότε έχω καλυφθεί στις ερωτήσεις. Ωραία. Ο κύριος Μωράης από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ελπίζω ότι ε, θα προλάβαινα να προετοιμάσω την δική μου ερώτηση όσο μιλούσε προλαλή σα, που ελπίζω ότι θα καθυστερούσε λίγο περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ τους δύο υπουργού, γιατί παρά τις πολιτικές μας διαφορές και θέσεις, σίγουρα αυτό το εξάμεινο ήταν πολύ έντονο από άποψη ε, συζητήσεων και προσπαθειών σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο τομείς. Ο πρώτος ενδιαφέρει άμεσα την ομάδα, πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας είπατε ότι κατά πάσα πιθανότητα το Συμβούλιο δεν θα ε, προλάβει, δεν θα είναι έτοιμο για να προωθήσει την οδηγία. Φαίνεται ότι μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του ανέλαβε και το Κοινοβούλιο τις ευθύνες του και ασχολήθηκε με το θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Εντολής για ποινικά ζητήματα εντολής προστασίας. Και όπως ξέρετε σήμερα ε, είχαμε και ψηφοφορία για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Γυναικών και στην ε, δική μας Επιτροπή προκειμένου να συνεχίσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Βέβαια, πολλές οργανώσεις πολιτών περιμένουν με υπομονησία το, την Ευρωπαϊκή Εντολή ε, Προστασίας και δεν θέλουν να καθυστερήσει εξαιτία ε, ε, ενδοκινοτικών διαφορών το θέμα. Γι' αυτό ήθελα να μας πείτε και τη δική σας γνώμη. Εμείς ευελπιστούσαμε ότι θα ευοδοθούν οι εργασίες και φαίνεται ότι καθυστερούν. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θα μιλήσουν για τη μετανάστευση σίγουρα και το άσυλο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό Πίτερ για το άσυλο που είπε ότι το πακέτο που ανεφέρθηκε στο πακέτο για το άσυλο Εκτιμούμε ιδιαίτερω ε, τι προσπάθειε σας, αλλά αυτό που προβληματίζει την ομάδα είναι ότι στο πακέτο για το άσυλο θέλουμε ποιοτική νομοθεσία μέχρι το 2012. Βέβαια, το 2012 είναι πολύ κοντά και όχι μόνο η δική σας Προεδρία, α, γιατί αυτό που θα πω δεν περιορίζει τη δική σα Προεδρία, πολλές Προεδρίες προσπάθησαν να προωθήσουν το πακέτο και εμείς θέλουμε ποιοτική νομοθεσία και για, τα, και για τη Eurodac, για τις διάφορες διαδικασίες. Σε ό,τι φορά το πακέτο της λάθρομετανάστευσης είναι πολύ ευαίσθητο, αλλά σημειώθηκε κάποιο πρόοδος και με αυτή την αισιόδοξη νότα θα ήθελα να ολοκληρώσω. Κυρία Βέμπερ από τους φιλελεύθερους, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο υπουργούς για την παρουσία τους και την παρουσίαση που μας έκαναν των συμπερασμάτων της Ουγγρικής Προεδρίας. Επικεντρώθηκαν κυρίως στα επιτεύγματα της Ουγγρικής Προεδρίας. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποιο προβληματισμό και ανησυχίες που έχουμε κατά το πέρας αυτής της Ουγγρικής Προεδρίας. Παρέμειναν αρκετές εκκρεμότητες, πολλά ανεπίλητα θέματα, οπότε αναρωτιόμαστε πώς θα τα χειριστεί η επερχόμενη Προεδρία και τι ε, κληροδότημα θα αφήσετε στην Πολωνική Προεδρία. Σε ό,τι αφορά την έκθεση Αντζελίλη και την προστασία των ανηλίκων, δυστυχώς ε, πολύ απέχουμε από την επίτευξη συμφωνίας και έχουμε αρκετά προβληματικά θέματα ε, φλέγοντα που θα πρέπει να συζητηθούν και θα περίμενα, θα ήλπιζα σε μεγαλύτερη ελαστικότητα του Συμβουλίου. Προηγουμένως αναφερθήκαμε και στο θέμα της ίσης ε, μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας, υπεπιθύσεων, ε, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσου προσανατολισμού και εκφράσαμε την απογοήτευσή μας για την αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων στη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε αμφίβολα στη Frontex, σε ό,τι αφορά το πακέτο του ασύλου, δυστυχώς έχουμε ακόμη πολλές ανησυχίες για το μέλλον. Και το, το, το Δουβλίνο 2 έμεινε τελείως απαράλλαχτο. Αναφέρθηκε και η κατάσταση στην Ελλάδα και φαίνεται ότι θα έπρεπε να είχε περιληφθεί και το Δουβλίνο 2. Σίγουρα η μετανάστευση και το άσυλο ήταν δύο τομείς που, που περιμέναμε πιο δραστήρια ανάμειξη και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολύ ασθενή της παρουσία μας απαγοήτευσε. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, θα έλεγα ότι και εκεί η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα ατυχής για την Ουγγρική Προεδρία, γιατί είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο, η Ουγγρική Προεδρία στο Συμβούλιο δεν μας βοήθησε για να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα. Το αντίθετο, αυτό που λάβαμε από την Εμπειρική Προεδρία είναι σημειώσεις, σημειώματα ότι μόνο οι πρόεδροι, οι σκιώδεις ηγητές και οι συντονιστές έχουν τέτοια πρόσβαση. Και χρειάστηκε πολύς χρόνος και οι βουλγαρικές και οι ρουμανικές αρχές είπαν ότι εκείνες τα πρόθυμες να επιτρέψουν πρόσβαση για να κατευνάσουν αυτή την θεσμική φιλονικία που είχαμε, τη διοργανική. Πώς πιστεύετε θα συνεχίσει η Πολωνική Προεδρία τις υποθέσεις αυτές. Για τους πρασίνους η κυρία Κέλλερ, ευχαριστώ. Όντως ήταν ε, πολύ φορτωμένο το εξάμεινο από άποψη εσωτερικών υποθέσεων και είδαμε πολλές προκλήσεις. Η μία ήταν η Σέγγεν και η δεύτερη ήταν η επαναστάση στη Βόρεια Αφρική. Για το Σέγγεν. Είδαμε ότι τα κράτη-μέλη διάλεγαν διάφορα σημεία από το πακέτο Σέγγεν και είχαμε πραγματικά μια τεράστια ευρωπαϊκή κρίση. Γιατί επλήγει μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν άκουσα τίποτα ούτε από το Συμβούλιο ούτε από την Προεδρία. Ε, τι γίνεται με αυτή τη διελκυστική και την προσπάθεια να αποδυναμωθεί το Σέγγεν. Το Συμβούλιο είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έπρεπε να υπεραμείνεται των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις επαναστάσεις στη Βόρεια Αφρική. Έχουμε δημοκρατικές επαναστάσεις εκεί. Οπότε κάποιος θα σκεφτόταν ότι η Προεδρία ή το Συμβούλιο θα καλωσόριζαν αυτές τις επαναστάσεις και θα, τις επαναστάσεις και θα στήριζαν αυτές τις χώρες στη δημοκρατική τους προσπάθεια. Αντίθετα, είδαμε μόνο το φόβο για την εισρωή των μεταναστών από τη Μεσόγειο και τι θα κάνουμε για να τους, μάλλον εις βάρος παρά για να τους προστατεύσουμε. Αυτό που θα περίμενα είναι προοδευτική δράση του Συμβουλίου και επιθυμία να βοηθήσουμε τις χώρες, το λαό τους, τους μετανάστες, καλύτερη υποδοχή των μεταναστών γιατί είχαμε 200 ε, που επαναγκαταστάθηκαν από την, ε, επαναπροωθήθηκαν από την ε, Μάλτα. Αλλά αυτό δεν ήταν καμία χειρονομία αυρότητας ή αλληλεγγύης. Δεν είχαμε καμία προσπάθεια επανεγκατάστασης μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική. Από ό,τι ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει προτάσεις που όμως δεν βρήκαν την υποστήριξη του Συμβουλίου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε την εμπειρία σας. Τι κάνατε για να προασπίσετε το Σέγγεν και τις θεμελιώδεις αξίες, τους μετανάστες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στις επαναστάσεις της Βορειοαφρικής. Εκ μέρους της Γκουα, κύριος Σταβάρας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επιδειξηγετικού ρόλου. Με το παράδειγμα, με την ικανότητα συντονισμού, με την ικανότητα υποβολής καινοτόμων ιδεών ή με την ικανότητα σωστής αντίδρασης στα γεγονότα. Από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι σε κανέναν από αυτούς τους τομείς ή με κανέναν από αυτούς τους τρόπους δεν ε, ε, πρωτοστάτησε η Ουγγαρία και πώς να πρωτοστατήσει εσωτερικές υποθέσεις και στη δικαιοσύνη αφού ε, με τον Ουγγρικό νόμο για τα μέσα μαζικής ενημέρωση, το Σύνταγμα το Ουγγρικό δεν, έδωσε, δεν είχε φοβερές επιδόσεις στο θέμα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, η Ουγγαρία. το Σέγγεν είναι σημαντικός πυλώνας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες και εκεί είχαμε πολλές εσωτερικές αντιπαραθέσεις στο Συμβούλιο και δυστυχώς η Ουγγαρία δεν κατάφερε να κατευνάσει αυτές τις διαφορές μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας και μετά με τη Δανία. Δεν κατάφερε να αντιδράσει ούτε στην κρίση της Βόρειας Αφρικής. Έμεινε και εκείνο το θέμα χωρίς καμία αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί διαπιστώσαμε ότι η σημαντικότερη πρόκληση που ανέκυψε για την Ουγγρική ε, Προεδρία στα μέσα της Προεδρίας δεν αντιμετωπίστηκε σωστά. Εγώ θεωρώ ότι μετά από πολύ έντονες πιέσεις ε, υπέβαλε τις προτάσεις της για τη μετακατάσταση των ε, μεταναστών, των προσφύγων η Ουγγρική Προεδρία. Περιμέναμε και η Ισπανία, ε, το Βέλγιο, η Ουγγαρία από τρεις προεδρίες περιμέναμε διακαώς την πρόταση. Τελικά ήρθε εμείς απαντήσαμε με αντιπρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέχρι στιγμής δεν έχουμε την αντίδραση της Ουγγρικής Προεδρίας σε σχέση με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσαν οι Υπουργοί σήμερα εδώ και τώρα να μας δώσουν μια απάντηση ως προς την αντιπρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι η συζήτηση θα διευκολυθεί και από το γεγονό ότι το ΕΛΚ απουσιάζει από τη συζήτηση. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει να πει τίποτα, είτε γιατί αποφεύγει την αξιολόγηση της Ουγγρικής Προεδρίας. Δεν έχει να πει τίποτα για αυτή. Ο κύριο Σόγκορ ε, έλαβε το λόγο εκ μέρου του ΕΛΚ και εκπροσώπησε το ΕΛΚ και μάλιστα πήρε το λόγο και πρώτο στο γύρο αυτό. Και μπορεί να μην εξάπλησε το χρόνο του, αλλά είχε τη διακριτική ευχαίρεια να μιλήσει όσο ήθελε. Ήταν ο πρώτο που έλαβε το λόγο ακριβώ γιατί εκπροσωπούσε το ΕΛΚ. Θα ακούσουμε τώρα το πρώτο γύρο απαντήσεων από τους δύο υπουργούς. Πρώτα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Ναυράτσης, που θα μας δώσει απαντήσεις. Ε, σας ευχαριστώ. Κύριε Μωράς, θα ήθελα πρώτα να απαντήσω στη δική σας ερώτηση, γιατί ε, ρωτήσατε για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία και αυτό ήταν σημαντικό στόχο και προτεραιότητα τη Ουγγρική Προεδρία. και επειδή η Βουλγική, η Ισπανική ε, και Ουγγρικοί Προεδρίες είχαν ε, αυτό το θέμα ως προτεραιότητα τους και από την αρχή είπαμε εμείς στην Ουγγρική Προεδρία ότι είναι κρίμα που δεν έχει σημειωθεί πρόοδος μέχρι τώρα, γι' αυτό και προωθήσαμε Θελήσαμε να δώσουμε νέα πνοή στην πρόταση αυτή και έτσι χειριστήκαμε και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία. Στις 18 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει το συνολικό πακέτο για την προστασία των θυμάτων που μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κύριο τμήματα. Το αναφορά την προστασία των θυμάτων αξιόπινων ε, πράξεων, εγκλημάτων και εκεί η Ουγγαρία υπέβαλε πολλές προτάσεις και υπάρχει και το πακέτο για την προστασία σε θέματα αστικού δικαίου. Βέβαια, ε, γνωρίζαμε αυτή εξ αρχής ότι η πρόοδος θα ήταν δυνατή μόνο αν καταφέρναμε συμφωνία για το διαχωρισμό του ποινικού από το σκέλος και την διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την ταχύτητα διεκπαιρέωσης τους. Βέβαια, στις αντίστοιχες ομάδες εργασίες, η πλειοψηφία των χωρών μελών θεώρησαν ότι είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι δύο τομείς, ώστε θα πρέπει να προωθούν και να εξεταστούν ταυτόχρονα. Γι' αυτό και ήταν πολύ αργή η πρόοδος. Πάντως, τουλάχιστον ξεπεράσαμε την αρχική αποτελμάτωση σε ό,τι αφορά αυτό το, την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Έχουμε τώρα στις ερωτήσεις κυρίας Βέμπερ για την προστασία των παιδιών κατά της ε, παιδικής παρογραφίας και κατά πολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Και εδώ μιλούμε για νέα μέτρα και σημειώσαμε τι πρόοδο. Είχαμε έξι τριμερείς διαλόγους στο τελευταίο εξάμεινο και πλησιάζουμε σε αίσιο πέρας των τριμερών αυτών διαλόγων. Βέβαια σε ορισμένους τομείς δεν έχει σημειωθεί εντυπωσιακή πρόοδος. Σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό των ιστοσελίδα που περιέχουν πορογραφικά στοιχεία ή την αφαίρεσή τους. Και το δεύτερο, ο δεύτερος τομέας αφορά το grooming. Δεν καταφέραμε να επιλύσω αυτά τα δύο θέματα στους τριμερείς διαλόγους, έχουν μείνει εκκρεμοί. Πάντως σε πολλούς τομείς πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο σε σχέση με την αρχική θέση. Τώρα Μα ζητήσατε να πείσουμε και τους ομολόγους μας στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά αν όντως επιτύχουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα θα έχουμε πιο εύκολη επίτευξη αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της, ε, των διακρίσεων. Αυτό εμπίπτει σε αρμοδιότητα άλλου συμβουλίου και δεν μπορώ να σας ενημερώσω για την πρόοδο ασχολείται με το θέμα αυτό η ΕΠΣΚΟ. Αυτά και νομίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις που είχαν απευθυνθεί σε μένα. κύριος Πίντερ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε γενικές γραμμές και ε, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις θα μπορούσα να πω το εξής μας προσάπτεται ότι η Ουγγρική Προεδρία δεν επέδειξε, λέτε, ηγετική στάση. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. 24 συμπεράσματα, 12 αποφάσεις του Συμβουλίου, ένας κανονισμός ή μία οδηγία εγκρίθηκαν. Εάν δούμε όλα αυτά τα στοιχεία, νομίζω μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι είχαμε μεγάλη αποφασιστικότητα Ιδιαίτερα δεν αν λάβουμε υπόψη, εκτός αυτού, ότι έχουμε και απόφαση ε, Συμβουλίου προσεχώς για τη σύμβαση του ΠΡΟΥΜ ή και μαζί με τη Frontex είναι τρία μόνο ε, τα ανοιχτά ζητήματα ε, τα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουμε μαζί σας. Και σε θέματα ε, παράνομης ε, και νόμιμης μετανάστευσης. Νομίζω εκεί πετύχαμε ως Προεδρία. Και νομίζω ότι μπορώ να πω ότι σε αυτό το εξάμεινο έγιναν ε, μεγάλες πρόοδοι. Ο κύριος Μωράες έχει δίκιο για το πακέτο του ασύλου. Πραγματικά χρειάζονται τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσουμε να, να εγκριθεί ε, πριν ε, λήξει η προθεσμία του προγράμματος της Στοχόλμης. Θα ήθελα να τονίσω ότι βεβαίως δεν έχουμε καταλήξει σε ό,τι αφορά την οδηγία για την άδεια παραμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα και κάτι ακόμα για την απασχόληση. Το επίζω να συμφωνήσουμε την άλλη εβδομάδα. Και σε ό,τι αφορά την οδηγία για την υποδοχή προσφύγων, στις 9 Ιουνίου άρχισαν οι συζητήσεις, αλλά το Συμβούλιο θα ασχοληθεί ουσιαστικά στη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου. Ο κανονισμός για τη Eurodac που ανέφερε και η κυρία Βέμπερ. 26 είναι τα κράτη-μέλη που επιθυμούν οι διοκτικές αρχές των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση ε, στη Eurodac, στην πρόσβαση δεδομένων για τις επανεγκαταστάσεις. Προσπαθήσαμε και με τους προκατόχους μας να συνεννοηθούμε για να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Πρέπει να σας πω ότι στο άσυλο νομίζω προχωρήσαμε πολύ ε, και πολλούς φακέλους προωθήσαμε, αλλά και τα άλλα θέματα που δεν έχουν λήξει νομίζω έχουν προετοιμαστεί ε, επαρκώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πω ακόμα το εξής στην κυρία Βέμπερ για το Σέγγεν. Γιατί μιλήσατε γι' αυτό. Δεν ήταν κρίση αυτό που έζησε το Συμβούλιο. Και δεν υφίσταται καμιά απειλή ε, για το Σέγγεν που είναι το μεγαλύτερο απίτευγμά μας. Έγιναν κάποιες νήξεις ε, κάτι υπενιγμή που αντιμετωπίσαμε, αλλά τίποτα που να απειλεί την ελευθερία ταξιδίων και διακίνησης και ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Το Συμβούλιο ενέκρινε μια σύσταση, στην κοινή απόφαση δηλαδή του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η Ρουμανία και η Βουλγαρία μπορούν να ενταχθούν στο Σέγγεν έτσι κι αλλιώ, το μόνο που εκκρεμεί είναι η ημερομηνία. Πότε θα ενταχθούν. Δηλαδή, βήματα έχουμε κάνει και εδώ. Θα ήθελα να πω το εξή στην κυρία Κέλλερ. Για το Σέγγεν. Το Συμβούλιο είχε μια ενιαία και στεναρή στάση την οποία υπερασπίστηκε με μεγάλη συνέπεια. Και για τη Βόρεια Αφρική. Κανένας πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχασε τη ζωή του στη Βόρεια Αφρική. Καταφέραμε να εκενώσουμε από τη Λιβύη όλους τους πολίτες της Ένωσης. Και σε σχέση με τα γεγονότα εκεί, η ύπατη εκπρόσωπος μετέβη στη Λιβύη όπως επίσης ε, και εκπρόσωποι ε, του κλάδου των εσωτερικών ε, υποθέσεων. Προσωπικά πήγα στη Μάλτα και λάβαμε από εκεί κάποια μέτρα. Και το κέντρο παρακολούθησης και ενημέρωσης, το ΜΙΚ, αμέσως ετέθησε λειτουργία, κινητοποιήθηκε και χάρη σε αυτά τα μέτρα δεν έχασε τη ζωή του, δεν απειλήθηκε κανένα πολίτη τη Ένωση. Και επίση δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι έχουμε 100 εκατομμύρια ευρώ ω χρηματοδοτικό μέσο ως χρηματική ενίσχυση που ε, απελευθερώθηκε αμέσως για τις χώρες που υφίστανται τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση. Βεβαίω και απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν στη Βόρεια Αφρική, αλίμονο. Αλλά αυτό δεν αφορά τα θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνη. Εκεί θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί το Συμβούλιο. Από τη Μάλτα εκενώθηκαν 1014 ακριβώς και 174 πολίτες του Τσάτ επέστρεψαν στην πατρίδα τους χάρη στη βοήθειά μας. Ενεστάλη και ε, το Δουβλίνο σε εκείνη την περίπτωση και ε, ε, έγινε ο επαναπατισμός. Έρχομαι τώρα στον κύριο Ταβάρες. Σας μίλησα για τα επιτεύγματα και για τις επιτυχίες που είχαμε. Ε, προφανώς για τις επιτυχίες θα σας μιλήσω. Ο καθένας εδώ ε, προτιμάει να μιλάει για τις επιτυχίες του. Υπάρχουν και κάποια αντιφατικά ε, και κάποιες αντιρρήσεις βέβαια. Δεν θέλω να παρουσιάσω την κατάσταση με τρόπο ιδιαίτερα ρόδινο, ιδιαίτερα απειλητικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Υπουργή. Θα ήθελα να πω στους υπουργούς της Ουγγρικής Προεδρίας ότι η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας συζητηθείτε και συζητείται εδώ στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Γυναικών. Σήμερα το πρωί είχαμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Γυναικών. Και τα μέλη και των δύο επιτροπών που συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση μου ανέθεσαν να απευθύνω επιστολή στην Προεδρία, την Ουγγρική προκειμένου, αλλά και στην επόμενη Πολωνική Προεδρία, όχι μόνο για να ενημερώσω ως προς την κατάσταση των πραγμάτων, αλλά για να τονίσω και τη σημασία που δίνεται σε αυτό το θέμα και από τις δύο αυτό το τόσο ευαίσθητο και λεπτό και σημαντικό θέμα. Είπαμε ότι είναι μείζον προτεραιότητά μας. η προστασία των ε, θυμάτων ε, εγκληματικών ε, ενεργειών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Ο κύριο Σόγκορ τώρα, που θέλει να ξαναπάρει το λόγο, δεν ξέρω ίσως για να απαντήσει σε κάποια θέματα που ακούστηκαν στις απαντήσεις. Επιτρέψτε μου να μιλήσω στα αγγουρικά. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ε, υποστηρίξω την Ουγγρική Προεδρία. Πολλές φορές έγινε λόγος για την υποστήριξη των ε, ΜΜΕ σε σχέση ε, με το θέμα του του συντονιστή όταν δεν είναι ο συνάδελφος από την ΙΝΚΟ. Spain, Hungarian and I'm... Όταν είναι εδώ ο κύριος Μπουσούτιλ από την ΙΝΚΟ, τότε εκπροσωπώ εγώ την ομάδα. Την ομάδα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά υποβλήθηκε δύο φορές μία ερώτηση προς, τα, προς εμένα και γι' αυτό έλαβα το λόγο δύο φορές. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως όταν η Ρουμανία το 2019 ε, εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα μπορέσω να υποβάλω την ερώτηση στα ρουμανικά. Στο μεταξύ μιλάω ουγγρικά και κάποια στιγμή μπορώ να λάβω στο λόγο και γερμανικά. Mr. member of this house. Ε, ευχαριστούμε κύριε Σόγκορ. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να εξηγεί γιατί εκφράζεται στη μία ή στην άλλη γλώσσα. Μπορείτε να εκφραστείτε σε όποια γλώσσα θέλετε. Στα αγγουρικά, ρουμανικά, όποια γλώσσα θέλετε. Πάντα είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας και μπορείτε να μιλήσετε είτε προσωπικά είτε εξ ονόματος της ε, ομάδας σας, κυρία Γκέντς. Και εγώ θα αρχίσω, συνεχίσω στα αγγουρικά, λέει η κυρία Γκέντς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας σήμερα το απόγευμα, γιατί πολλά ελέγχθησαν για το Σέγγεν, που είναι μία από τις βασικότερες προκλήσεις της Ουγγρικής Προεδρίας. Και χαίρομαι γιατί η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα προσχωρήσουν στο χώρο του Σέγγεν. Υπήρξαν πολλές προσδοκίες οι οποίες εκφράστηκαν και χαίρομαι για τα πράγματα κινήθηκαν στο μεταξύ. Μία ε, επιπρόσθετη ερώτηση θα ήθελα να υποβάλω. Η Ουγγρική κυβέρνηση βοήθησε ετούντες ασύλο. Αυτό σημαίνει ότι ε, μετέβησαν εκεί πρόσφυγες ή μετανάστες διότι έφτασαν στη Λαμπετούζα και στη Μάλτα ε, πάρα πολύ και νομίζω ότι ο αριθμός των 200 που ανέλαβαν ορισμένε χώρες είναι πολύ μικρός αριθμός. Ποιο ρόλο διαδραμάτισε η ε, Ουγγαρία. Κύριε Ναυρατζής, τι γίνεται σε σχέση με την, ο... την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων, διότι εμεί θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει επί του θέματος. Μιλήσαμε για την στρατηγική υπέρ των Ρωμά, που είναι μία από τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με το Ουγγρικό Σύνταγμα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο φτάσαμε σε αυτά συμπεράσματα ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως προβαίνει σε αποτιμήσεις, αλλά η Ουγγαρία δεν λάμπει δια της παρουσίας της σε αυτό το τομέα. Εσείς είσαστε αναπληρωτής Πρωθυπουργό και Υπουργός Δικαιοσύνης και νομίζω ότι φέρετε μεγάλη ευθύνη για την ποιότητα της νομοθεσίας που είναι απότοκη του συντάγματος. Ποιοι μηχανισμοί προβλέπονται μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, θεσμοθέτησης. Θα πρέπει να μιλάμε για τα δικαιώματα των πολιτών και να τα υπερασπιζόμαστε. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, αλλά πέρα από τα πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα που όλοι αναγνωρίζουμε, τι κάνατε ως προς τον νόμο των ΜΜΕ, διότι από όσο γνωρίζω, στο τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας θα ανακύψει ένα άλλο ψήφισμα του Κοινοβουλίου και έχει μεγάλη σημασία τι έχετε επιτύχει επί του θέματος. Αναρωτιέμαι αν έχει επιτελεστεί κάποια ε, πρόοδος επί του θέματος. Τι έχει γίνει σε σχέση με τις εξελίξεις του συντάγματος Φίξτρομ και εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου. Έχουμε μπροστά μας την προθεσμία του 2012. Εγώ είμαι εισηγήτρια για τον κανονισμό 2 του Δουβλίνου. Και για να είμαι ειλικρινής, είχα πολύ υψηλέ προσδοκίε από την Ουγγρική Προεδρία, ότι δηλαδή θα μπορούσατε να άρετε το αδιέξοδο, διότι αυτό είναι και ο στυλοβάτης του συστήματος ε, χορήγησης ασύλου. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας. Είσαστε ικανοποιημένοι με την ε, πρόοδο του πακέτου χορήγησης ασύλου και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των νέων οδηγιών ε, αποδοχής σε σχέση δηλαδή με την οδηγία περί υποδοχής ε, τούντων άσυλο θεωρείτε ότι έχουμε να προσμένουμε κάτι από εσά από τη μελλοντική Προεδρία έτσι ώστε να άρουμε αυτό το ε, αδιέξοδο και να αρχίσουμε το τριμερή διάλογο σε αυτό το βασικό θέμα. Η κυρία Ζίμπελ. Όχι. Η κυρία Γκυγιόν. Ευχαριστώ. Μέσα στα πλαίσια αυτής της, αυτού του απολογισμού της Προεδρίας θα ήθελα να σταθούμε σε θέματα ασύλου. Μιλήσατε για πρόοδο. Αλλά έχει σημασία να δούμε ποια είναι τα μικρά βήματα που επιτυγχάνονται. Δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας ως προς την, ε, την πρόοδο. Θα δούμε κατά πώς έχει επιτελεστεί πρόοδος ως προς την οικογένεια, τον ορισμό της οικογένειας και ούτω καθεξής. Επίσης μιλήσατε για το πακέτο ασύλου για το 2012, το οποίο θα ολοκληρωθεί πολλά κείμενα όμως του πακέτου ε, αφισβητούνται, δηλαδή δεν έχει επιτελεστεί η απαιτούμενη πρόοδος ως προς τις νέες προτάσεις υποδοχής ε, θα ήθελα να εκφέρω πολλές επιφυλάξεις και είχαμε και πολλές απορρίψεις από τα κράτη-μέλη, μην το ξεχνάμε αυτό. Θα μπορέσετε να μου μεταβιβάσετε ένα μέρος της αισιοδοξία σας για το μέλλον. Η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Ουγγρική Πρόεδρη είχε να αντιμετωπίσει μία ε, ιδιαίτερα δυσχερή περίοδο ε, για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Ήδη δεν είναι εύκολος ο τομέας ε, αυτού. Γιατί πάντα πρέπει να γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι. Αλλά ως προς τα θέματα της μετανάστευσης, του Σέγγεν και του Σέγγεν ιδιαίτερα, αντιμετωπίσαμε πολλά. Όμως είναι ιδιαίτερα ατυχές το γεγονός των τεκτενόμενων στη Βουδαπέστη, κάτι το οποίο δυσχέρανε το έργο της Ουγγρικής Προεδρίας. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ επί του θέματος. Ίσως αποκλίνουν οι απόψεις μας. Έγιναν ζωηρές συζητήσεις για το Σύνταγμα, για το νόμο περί ΜΜΕ, αλλά το θέμα του χρονισμού ήταν πολύ δύσκολο και εν πάση περιπτώσει δεν είχατε να επιδείξετε και λαμπρό έργο ως προς τα μέτρα που λάβατε στο τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν καθόλου ε, εύκολο αυτό το πακέτο. Όμως έγινε πρόοδος σε άλλα θέματα. Στο, στην επιστολή δικαιωμάτων με την κυρία Σίμπελ το είδαμε αυτό το θέμα. Βλέπουμε πώς, έχει, πώς σκιαγραφείται το θέμα και η συμφωνία και ελπίζω να κλείσει σύντομα. Ε, όχι ίσως υπό Ουγγρική Προεδρία, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς θα έχετε διεκπαιρεώσει το μεγαλύτερο ε, μέρος ε, του έργου, όπως μας είχε πει και ο κύριος ε, Ζάνκερ. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα ήδη έχει διεκπαιρεωθεί εμπολής. Είναι πολύ κρίμα γιατί η Προεδρία σας δεν πρόθυσε το θέμα για την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον χώρο Σέγγεν. Γιατί τώρα θα γίνει η νέα αξιολόγηση Σέγγεν και ίσως υπάρξει σύμπτωση των δύο. Δεν το διεκπαιρεώσατε το θέμα. Και αυτό δεν πρέπει να το συγχαίουμε με το θέμα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας που πληρούν τα κριτήρια προσχώρησης. Επίσης δεν συμμερίζομαι τη θέση του κυρίου Πίντερ περί προσπέλασης στα στοιχεία της Eurodac. Πρόκειται για κάτι πολύ δύσκολο και δεν θα διεκπαιρεωθεί τόσο εύκολα στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ. Όπως είπα και προηγουμένως, στις 4.30 έχουμε προγραμματίσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι χρειάζεται τις ηλεκτρονικές σας κάρτες και αν τις έχετε ξεχάσει στείλτε κάποιον να σας τις φέρει. Γιατί με το που θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος γύρος των απαντήσεων από τους δύο υπουργούς θα περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Υπάρχει και άλλη ερώτηση. Δεν σας είχα σημειώσει. Είστε ο τελευταίος ομιλητής, αλλά παρακαλώ χρόνου φίδου, ώστε να προλάβουν και οι δύο υπουργοί να μιλήσουν από ένα πεντάλεπτο. Αναφέρθηκε η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η εφαρμογή της. Αναφέρθηκε δεν υπάρχουν προβλήματα με το χάρτη αυτό, ότι είναι συνεπής, συμπληρωματικός κτλ. Κάτι που δεν ακούστηκε στη γενική συζήτηση είναι η πιθανότητα ε, διαμάχης μεταξύ αντικρώμενων συμφερόντων, μεταξύ κάποιων δικαιωμάτων του χάρτη ή ε, μεταξύ του χάρτη και του, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης. Φαίνεται ότι εκεί έχουν χαθεί κάποια δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά τις θρησκείες, φαίνεται ότι υπάρχει ισότητα μεταξύ ορισμένων θρησκειών και όχι μεταξύ όλων των θρησκειών. Στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο ορισμένοι ε, ε, γιατροί δεν δικαιούνται να δηλώνουν ότι είναι, χριστιανοί, ότι είναι χριστιανοί, κάτι που δεν ισχύει για τα άλλα επαγγέλματα. Φαίνεται ότι ανεξιθρησκεία διεκδικείται για ορισμένε μόνο θρησκείες. Νομίζω ότι μερικές φορές ε, η πράσπιση των ε, ε, ορισμένων δικαιωμάτων γίνεται με επίκληση συναισθηματικών περισσότερο και συγκινησιακά φορτισμένων επιχειρημάτων. Κατά τη γνώμη μου, τα, το θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης εκλογών του συνεταιρίζεσθε θα πρέπει να υπερισχύουν ε, από, τη, από άλλα, να υπερισχύουν άλλων δικαιωμάτων. Ε, το δικαίωμα να προσβάλλει κάποιος για παράδειγμα. Νομίζω ότι ε, προτιμώ να λέω ελεύθερα αυτά που πιστεύω παρά να περιορίζω την ελευθερία έκφραση του άλλου. Επίσης θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο κοινό ότι μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ της συλλογική κριτικής και της παράλογης κριτικής. Ευχαριστούμε κύριε Μπρος. Θα δώσουμε τώρα από ένα πεντάλεπτο στον κάθε υπουργό για να απαντήσει. Πρώτα ο Υπουργός Ναυράτσιτς. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται καν να εξαντλήσω το πεντάλεπτο. Να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Γκέντς για την οριζόντια οδηγία καταπολέμησης ε, των διακρίσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω, εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΠΣΚΟ και όχι στο Συμβούλιο ε, Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης. Δεν μπορώ να σας ενημερώσω για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Κυρία Λάτφορτ, θέσετε μία ερώτηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων και τη συζήτηση για το νόμο περί μη ε, που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες στην Ουγγαρία. Μετά από το πρώτο εξάμεινο συζητήσεων φαίνεται ότι οι φόβοι που αρχικά είχαν διατυπωθεί το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο κατά της νομοθεσίας ε, στην Ουγγαρία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φαίνεται ότι είναι αβάσιμη όλη αυτή η φόβη. Αποδείχθηκαν τελείως ανυπόστατοι γιατί πραγματικά υπάρχει ελευθερία με μία ε στην Ουγγαρία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι φυσταθούν πια αυτά τα επιχειρήματα. Τώρα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος, και πάλι το θέμα του συγχρονισμού δεν είναι και πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι η στιγμή της υποβολής αναθεώρησης, αλλά το κατά πόσο καλό είναι το Σύνταγμα. Αυτό διαφέρει περισσότερο παρά η χρονική στιγμή της αναθεώρησης. Γιατί όταν είναι πρόσφορες οι συνθήκες και όταν υπάρχει ε, η απαιτούμενη πλειοψηφία, τότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υποβολή και των προτάσεων για αναθεώρηση του συντάγματο. Σίγουρα υπάρχει, κύριε Μπρόγκ, μια διαμάχη μεταξύ ε, συμφερών, ε, ε, δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μερικές φορές υπάρχουν αντικρουόμενα δικαιώματα και υπάρχουν και χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ισχυρότερο και πιο μικροχρόνιο δημοκρατικό παρελθόν. Άλλες χώρες όμως που μόλις πριν από 20 χρόνια ανέκτησαν την ανεξαρτησία τους και αποτείναξαν έναν απολυταρχικό και δικτατορικό ζυγό για αυτές, το γεγονός ότι υπάρχει ένας μηχανισμός, εγκυμένος μηχανισμός προστασίας των θεμελιδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά ε, υπερτερεί το κοινοτικό σύστημα κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με τις εθνικές. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάνουμε απολογισμό της Ουγγρικής Προεδρίας. Παρακαλώ λοιπόν ησυχία στην αίθουσα για να ακούσουμε και τους δύο υπουργούς. Κύριε Πίντερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα και τηλεγραφικά, γιατί έχουμε και τη χρονική αυτή πίεση. Ε, να απαντήσω το εξής πρώτα απ' όλα στην κυρία Γκιόνς δεν πρόκειται για 200. 1014 σας είπα κατάφεραν να γίνουν δεκτοί στη Μάλτα. Και 174 ήταν οι πολίτες του Τσάτ που κατάφεραν να επαναπροωθηθούν. Αφήστε δε που προηγουμένως είχαν φτάσει στη Μάλτα άλλες 5.000 πρόσφυγες. Και καμία άλλη προεδρία δεν είχε αποπειραθεί να ε, ελαφρύνει λίγο την πίεση που δέχεται αυτή τη αφόρητη η ε, Μάλτα. Μόνο η Ουγγρική Προεδρία εισάκουσε τις ε, φωνές της Μάλτας που ζητούσε βοήθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2, η κατάσταση είναι λίγο πατ με όρους κακιού. Είναι δύσκολο γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η μεταναστευτική πίεση. Στο παρελθόν αυτό φορούσε μόνο την Ελλάδα, τώρα έχουμε τη Μάλτα, την Ιταλία και σιγά σιγά θα έρθει και η ώρα της Γαλλίας. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει ο κανονισμός του Δουβλίνου. Ε, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα αυτό το θέμα. Μιλήσατε επίσης για την οδηγία ε, και τις ε, διαδικασίες και τα σχέδια για την υποδοχή προσφύγων ε, ετών των Υπάρχουν διάφορα σχέδια, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση. Στις 19 ε, άρχισε πολύ πρόσφατα να εργάζεται ο αντίστοιχο οργανισμός στην Ελλάδα και σας είπα για τον κανονισμό του Eurodac, 26 είναι τα κράτη-μέλη που συμφώνησαν και ζητούν να έχουν πρόσβαση ιδιοκτικές τους αρχές ε, στη βάση δεδομένων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται ε, για την ασφάλεια όλων μας και στο μέλλον. Για τη δέσμη για το άσυλο και την προθεσμία του 2012 νομίζουμε ότι μπορεί να τηρηθεί εάν λύσει τρία θέματα κάθε Προεδρία και αν εργαστούν με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς και οι τρεις επόμενες Προεδρίες. Είμαι βέβαιος ότι θα τηρήσουμε αυτές τις προθεσμίες. Κυρία Λάτφορτ. Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολη η καιρή ε, και ακριβώς σε τέτοιους καιρούς ε, φαίνεται που είναι το σύνορο ανάμεσα στο εφικτό και το ανέφικτο της πολιτικής. Σε ό,τι αφορά ε, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου εγκρίθηκαν, δηλαδή έχει αποφανθεί το Συμβούλιο. Και δεν μπορούν πλέον ε, να προκύψουν νέοι όροι και προϋποθέσεις για τις δύο αυτές χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για την υποστήριξή σας. Thank you, thank you. We thank both... Ευχαριστώ. ευχαριστούμε και τους δύο υπουργούς και το επιτελείο τους ε, για τις εργασίες του εξαμήνου. Ε, τους ευχόμαστε καλή λήξη, καλό υπόλοιπο της Ουγγρικής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ. Σκεφτείτε και το χρόνο. Είχαμε πει ότι θα ψηφίσουμε στις 4.30. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρούμε το χρονοδιάγραμμά μας. Hello? Again, again colleagues. Λοιπόν, συνάδελφοι, θυμίζω πάλι πόσο σημαντικό είναι να έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες έτοιμες. Is anyone aware of the voting card thing? Τα ξέρετε όλα αυτά τα περί κάρτας και πώς ψηφίζουμε. No one is having a problem with the electronic card. Είμαστε όλοι εντάξει, έχει κανείς πρόβλημα με την ηλεκτρονική του κάρτα. Ε, ναι, η κυρία Χάουταλα. Είναι σκάνδαλο, η ίδια η συγκήτρια δεν έχει κάρτα, αλλά έχω στείλει να μου τη φέρουνε. Εντάξει, ωραία, κάτι κάνατε ήδη, έχετε στείλει, προς το παρόν θα ψηφίσετε. Α, να περιμένουμε μια στιγμή τότε. Είναι καθοδόν η κάρτα σας από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα. Εντάξει, κυρία Χάουταλα. Ναι, ντρέπομαι πάρα πολύ, αλλά θα χρειαστούν 6-7 λεπτά. Και δεν θα τολμούσα να χάσουμε τόσο πολύ χρόνο όλοι μαζί. Ε, αν μου επιτρέπετε θα σηκώνω το χέρι μου. Εντάξει, για την πρώτη ψηφοφορία θα σας λαμβάνουμε υπόψη. Έτσι. Θα μας σηκώνετε το χέρι σας και θα μετράμε. Χειροποίητα be getting started. We have, if I'm not mistaken, five electronic... Αν δεν απατώμε έχουμε πέντε ηλεκτρονικέ ψηφοφορίε. Λοιπόν, πάμε στο 12. 13, 14 και πάει λέγοντα, 15 και 16. Το πρώτο θέμα είναι τι έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα έγκριση του σχεδίου έκθεση. Η συγκίτρια είναι η συνάδελφο κυρία Χαουταλά, αυτοπροσώπο, το 13 φορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Αυστραλία. Α, όχι. Το 13 δεν θα ψηφιστεί, έχει καταργηθεί. 14. Αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις. είναι Τβέλ την εισηγήτρια. 15 συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εισήγητη ο κύριος Αξιλφό. Και το 16 είναι η υπηρεσία για την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων προφόρηση μεγάλη κλίμακα στον τομέα ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Έγκριση και δύο εκθέσεω. Εισηγητή ο κύριο Κάρλο Κοέλιο. Εντάξει είμαστε. Αρχίζουμε από το 12, η κυρία Χάουταλα, ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι το σημείο 13 της κυρίας Σινετβέλτ δεν θα ψηφιστεί σήμερα. Ναι. Έτσι όπως λέει η μερίσια διάταξη, που κρατάω στα χέρια μου, το σημείο 13 που αφορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για το PNR, τα δεδομένα των καταστάσεων επιβατών, έχει αποσυρθεί από την ημέρη διάταξη. Δεν θα εγκριθεί. Έχει βγει Το 14 είναι επίση τη κυρία Σινετφέλτ. Αλλά είναι άλλο θέμα. Α, μάλιστα, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, κύριε Πρόεδρε. So, we are getting started by point... Αρχίζουμε με το 12, όπως είπαμε. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Η συγγήτρια. Η κυρία Χάουταλα. Θα τη μετράτε. Όταν σηκώνει το χέρι της. Γιατί δεν, έφτασε ακόμα η κάρτα. Πάμε. Η τροπολογία υπαριθμό 18. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. Ψήφι υπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος. Γι' αυτό τις έχουμε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και κάρτες. Αρχίζει παρακαλώ η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρασε. 25 κατά, 21 υπέρ, απορρίπτεται. Τμήμα δεύτερο. Ψήφι υπέρ. Against, abstentions, adopted. Κατά υπέρ εγκρίνει. Αποχές εγκρίνεται, συγγνώμη. 19 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 20. Υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 21. Υπέ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Παρακαλώ. Για την 21. Την 21 ελέγχουμε. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει. «25 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται». Δεν πειράζει όποιος φυλάει τα ρόχα του. Ε, συμβαστική 2. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπέρ 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Όχι, 28 επέζησε, λέει ο πρόεδρος. Ψήφι υπέρ 28. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Για την 29 παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα. Πέρασε. 24 υπέρ, 22 κατά εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τριάντα επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 35 πρέπει να την ψηφίσουμε, γιατί υπήρξε συμβαστική εκεί. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα Πού πάμε? Στη συμβιβαστική υπαριθμό 6. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο θέλετε. Ελέγχουμε την 53 λοιπόν. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική υπολήθευση. Πέρασε. Yes, rejected. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η βαστική 7 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Η βαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 60 Επέ. κατά αποχές απορρίπτεται 61 είπε. κατά αποχές απορρίπτεται 62 με προφορική της εισηγήτριας είπε. κατά αποχές εγκρίνεται 26 παραγραφούς με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην νέα συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον. Υπέρ Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 69. Παρακαλώ αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Ω, λυπάμαι πολύ, συγγνώμη. Και ερχόμαστε τότε στη συμβαστική 11. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71. Favor. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 προφορική των φιλελευθέρων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατά τμήματα ή 82. Τμήμα πρώτον. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε τις 82. Ηλεκτρονικά αρχης τώρα ψηφοφορία. Πέρας. 26-21 εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Amendment 83. Favor. 83 υπέρ. Κατά. Το ξέχασα. 39. Με προφορική τροπολογία της εισηγήτρες. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83, πάντα στην παράγραφο 39, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα το 84. Κατά τμήματα με προφορική τροπολογία τμήμα πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 κατά τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ Against. κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Οι σκέψη σκέψεις τώρα. Η τροπολογία 1, υπέρ. Against, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 5, κατά τμήματα, τμήμα πρώτο, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, η τροπολογία 7 υπέρ, κατά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 Κάτι μου λένε ότι ξεχάσαμε να ψηφίσουμε τη 37. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Λυπάμαι πάρα πολύ. 37. Στη σελίδα 3 είναι το καταλόγο ψηφοφορία. Μου λένε ότι ξεχάσαμε την ψηφίσουμε αυτή. Κάναμε τέτοιο πράγμα. Ε, μπορούμε να την ψηφίσουμε. Στη σελίδα 3. Ψήφι υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Όχι υπέρ, είναι ηλεκτρονικό αυτό. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε η τελική ψηφοφορία αρχίζει τώρα παρακαλώ. Πέρας. 47 υπέρ, 2 κατά συγχαρητήρια κυρία Χάουταλα. Now. Now. Προχωράμε στην επόμενη ψηφοφορία. κύριε Αντιβέλτ. Κύριε Πρόεδρε, με κάποιες επιφυλάξεις θα πρότεινα αναβολή της ψηφοφορίας ε, της έκθεσής μου, γιατί βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για συμβαστικές λύσεις ε, εγώ θεώρησα ότι το πακέτο των συμβαστικών λύσεων ήταν όριμο για την ψηφοφορία, αλλά πριν από λίγο μία ομάδα μου ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να υποστηρίξει τις συμβαστικές προτάσεις με τη μορφή που έχουν τώρα, δεδομένη της σημασίας τους και της σπουδαιότητας του θέματος, περι, προτιμώ να περιμένουμε λίγο ακόμη, αναβάλλοντας την ψηφοφορία, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πακέτο που θα τη χάνει ευρεία συμφωνίας. Καλώς. Νομίζω ότι μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση της συγγετρίας κυρίας Εντφέλτ. Οπότε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, συμφωνούμε μαζί της για αναβολή της ψηφοφορίας. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Μία διευκρίνηση. Μία από τις ομάδες πιστεύει ότι δεν ε, ε, ακούστηκε δεόντως η άποψή της για τις συμβαστικές προτάσεις. Συμφωνούμε με τις περισσότερες από αυτές, αλλά λυπόμαστε γιατί οι περισσότερες από τις πολυάριθμες τροπολογίες που κατατέθηκαν για την πολύ αυτή σημαντική έκθεση αγνοήθηκαν στη διάρκεια των διπραγματεύσεων για την ανέβρεση συμβαστικών λύσεων. Και είμαστε ε, απρόθυμοι, αλλά παρόλα αυτά θα συμφωνήσουμε με την αναβολή ευελπιστώντα ότι θα έχουμε καλύτερη συνεργασία με την εισηγήτρια στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Με βαριά καρδιά συμφωνούμε με την αναβολή. Ο κύριος Μωράης. Προσπάθησα να ψηφίσω την άνοιξη στο μικρόφωνο, συμφωνώ και εγώ πάντως με την αναβολή. Οκ, okay. η κυρία Βίμπερ, κύριος... Κύρκοφ. Και εμείς φιλελεύθεροι είμαστε, η συγκέντριά μας φιλελεύθερη είναι, κανένα πρόβλημα. Κύρκοφ, συμφωνώ. Αλλά θα προτιμούσα να είχαμε συνεννοηθεί προηγουμένως, να είχε ζητηθεί και η δική μας γνώμη. Επειδή κανένας ρώτησε τη γνώμη μας, κανονικά θα ήμουν κατά της αναβολής. Παρ' όλα αυτά Έστω και με βαριά καρδιά, συμφωνώ με το αίτημα αναβολή, ευελπιστώντα ότι θα καταλήξουμε τελικά σε συμφωνία για τι συμβαστικέ λύσει. Εμεί μέχρι στιγμή είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μα με την εισηγήτρια. Σεβόμαστε την επιθυμία μας, την επιθυμία της και συμφωνούμε με την πρόταση αναβόλης. Ο κύριος Μποργέτζο και εμείς είμαστε υπέρ της αναβόλης. Σαρτζεντίνη για τους πράσινους. φαίνεται ότι έχει συγκεντρωθεί πλειοψηφία για την αναβολή. Εντάξει. Ε, θα το δεχτούμε και αυτό. Πάντως υπήρχε ήδη διαμορφωμένη συμβαστική πρόταση. Ήμασταν έτοιμοι να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω προς τι αναβολή. Εμείς δεν ε, είμαστε υπέρ μιας νέας χρονοβόρας διαδικασίας. Ναι, αλλά υπευλήθη πρόταση από την εισηγήτρια και στόχος ακριβώς είναι να εξασφαλίσει λίγο χρόνο προκειμένου να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις και να συγκεντρωθεί όλο και μεγαλύτερη συνένεση από τις ομάδες. ώστε πραγματικά να ψηφίσουν με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Κυρία εισηγητρία, κυρία Αντφέλτ, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους και άκουσα και κατανόησα το σχόλιο του κ. Κύρφου. Δεν ήταν δική μου αυτή η ιδέα αρχικά και σε καμία περίπτωση θα το πρότεινα αν δεν το έκρινα απαραίτητο. Και πραγματικά είναι ατυχέ ε, που πήραν τέτοια τροπή τα πράγματα. Φυσικά όλοι συμμετέχουμε στην πραγματεύση καλή την πίστη και όταν καταλήγουμε συμβαστικέ ε, προτάσει θεωρούμε ότι υπάρχει συνένεση και τι ασθενίζονται όλοι. Εν πάση περιπτώσει είναι έκθεση πρωτοβουλία, δεν είναι νομοθετική έκθεση. Οπότε, αν υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε σε πρόταση κοινή αποδοχή, γιατί να μην το επιχειρήσουμε. Καλώ, οι συντονιστέ συμφώνησαν με την αναβολή. Βλέπω όμω ότι ο κύριο Δία Δεμέδα και η κυρία Χιμένε ζήτησαν το λόγο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, φυσικά και θέλω να προσθέσω. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι δέχομαι την απόφαση της πολιτικής μου ομάδας φυσικά και αποδέχομαι την πρόταση της πολιτικής μου να δεχτούμε την αναβολή. Αλλά δεν θα ήμουν, δεν θα είχα τη συνείδησή μου αν δεν σας εξέφραζα και την γνώμη μου. Εγώ κατέθεσα 38 τροπολογίες για την έκθεση και ούτε μία φορά δεν ζήτησε τη γνώμη μου η συγγήτρια. Η συγγήτρια δεν μου τηλεφώνησε ούτε μία φορά για να συνομιλήσουμε και να αναλύσουμε καμία από τις, ε, οποιαδήποτε από τις 38 μου τροπολογίες. Και εγώ δεν κάνω τον σκιώδη εισηγητή της ομάδας. Έχω, έχουμε την Άνια Χάρκης που είναι σκιώδη εισηγητρία και ε, δέχομαι τις προτάσεις Αλλά για τις δικές μου τροπολογίες υπεύθυνο είμαι εγώ και τις κατέθεσα από κοινού με τον κύριο Λουίς Δεγκράντες. Και για τις τροπολογίες αυτές αρμόδιοι είμαστε εμείς. Και θα προτιμούσαμε ως, ως τροπολογιών είχαμε ε, συμμετέχει, να είχαμε λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις και να βρούμε κάποια σημεία ε, συμφωνίας ή να εντοπίσουμε τις διαφωνίες. Μέχρι πριν από λίγο όμως καμία χειρονομία επικοινωνίας, η διάθεση ομως καμια χειρονομια επικοινωνία, η διαθεση επικοινωνιας δεν έδειξε συγκεντρία απέναντί μου. Σέβομαι μεν την ε, πρόταση της ομάδας, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτα δικαιολόγητη αυτή η αναβολή τη ψηφοφορία. Οκ, αλλά εμείς αποφασίσαμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία γιατί όλοι οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούν τις ομάδες τους συμφώνησαν με την αναβολή. Αλλά ζήτησε κάποιο κάποιος επιπλέον το λόγο και το θεώρησα σκόπιμο να σας δώσουμε το λόγο κύριε Δίας Δεμέρα. Ας ακούσουμε και την εισηγητριά σας, την κυρία Χάνκης, αλλά ζήτησε το λόγο προηγουμένως και η κυρία Χιμένες. Μια στιγμή κυρία Χάνκινς. Πρώτα η κυρία Χιμένες Μπεσερίλ και μετά εσείς. Δύο λόγια μόνο. Συμφωνώ με τον κύριο Διαστεμέρα. Γιατί και εγώ κατέθεσα 14 στον αριθμό για τα θύματα της τρομοκρατίας. Και εδώ και χρόνια ασχολούμαι με θύματα της τρομοκρατίας και είμαι και εγώ προσωπικά θύμα της τρομοκρατίας. Και Μέχρι στιγμής έλαβα μόνο μία μικρή συμβαστική πρόταση που απέκλειε ούτως ή άλλως τις δικές μου τροπολογίες. ασχολήθηκα και με άλλε εκθέσει, όπω την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία των Θυμάτων. Και είχαμε μακροχρόνιε διαπραγματεύσει και είχα πολλέ συνομιλίε με του συντάκτε των τροπολογιών. Στην περίπτωση αυτή, η συγγήτρια, όπω είπε ο κύριο Δία Δεμέρα για τι δικέ του 40 τροπολογίε με τον κύριο Δεγκράντε Πασκουάλ, εμεί αγνοηθήκαμε. Η εισηγήτρια μα αγνώρισε, δεν μα εμπεριέλαβε καθόλου στι διαπραγματεύσει. Εγώ είμαι κατά τη αναβολή. Κυρία Χάνκη, Θέλετε το λόγο ως κοιόδηση συγγήτρια του ΕΛΚ για την έκθεση Εντβέλτ. Θα μιλήσω ογκρικά κύριε Πρόεδρε, γιατί το πρόβλημα που είχαμε σε προηγούμενη συζήτηση ήταν ότι μιλούσα αγγλικά. Και ελπίζω να γίνω καλύτερα κατανοητή μιλώντας τη μητρική μου γλώσσα. Εγώ είμαι η σκιώδη του ΕΛΚ και πιστεύω ότι η ομάδα μας υιοθέτησε μια πολύ σωστή θέση. Είχαμε πολλές συναντήσεις και άτυπες και νομίζω ότι εκεί αποσαφηνίστηκε η θέση μας. Νομίζω ότι ε, διευκρίνησα πλήρως τη θέση του ΕΛ και τη δική μου ως και οδουσικητρίας. Το μείζον ζήτημα εδώ δεν είναι κάτι που αφορά την πολιτική πρακτική, αφορά θέματα αρχής. Δεν μπορούμε να αντιστρατευόμαστε τέτοιες αρχές, γιατί έτσι είμαστε ασυνεπείς ως προς τις αξίες μας. Και σε ό,τι αφορά τις 19 βασικές τροπολογίες, βασικές ε, ψηφοφορίες, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την ε, βασική θέση του ΕΛΚ όσο και αν χρονοτριβούμε, η θέση μας δεν θα αλλάξει ως προς τις 19 ε, νευραλγικές ψηφοφορίες για μας. Δεν νομίζω ότι η περαιτέρω χρονοτριβή καθυστέρηση θα βοηθήσει, γιατί δεν νομίζω ότι θα συγκαλυφθούν ή θα απαλληθούν οι διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν για την αναβολή. Αυτό το αποφασίσαμε λοιπόν. Δεν χρειάζεται να επανέλθουμε στο θέμα επί της ουσίας ή κατά πόσο είναι σκόπιμη η αναβολή. Ακριβώς ε, για να διευρυνθεί, να πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες ανέβρεσης συμβαστικής λύσης, παρατείνουμε λίγο το χρόνο για τις διαπραγματεύσεις. Μετά από αίτημα της συγκεντρία. Η κυρία Έντβελτ έχει πάλι το λόγο. Πραγματικά είναι ατυχή αυτή η κατάσταση και να διορθώσω μια παρεξήγηση. Είχα διαβουλεύσεις με Ισπανούς ευρωβουλευτές και έχουμε, έχω και γραπτές αποδείξεις, έχω τα mail που σας έστειλα και σε εσά κύριε Δίας, γιατί εγώ προσωπικά έγραψα το mail, όχι βοηθός μου. Και σας υπέβαλα προτάσεις, μπορεί να μην τις δεχτήκατε, αλλά μην μου λέτε ότι δεν είχα επαφή με κανέναν, ότι σας αγνόησα. Έχουμε ένα σύστημα στο Κοινοβούλιο με σκιώδεις συγητές. Οποιοςδήποτε μπορεί να καταθέσει τροπολογία, αλλά ε, εφόσον δεν τις εστερνιστεί, δεν τις παρουσιάσει ε, παρκώς ο σκιώδης συγητής, μπορεί να μην ληφθούν υπόψη. Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα, είναι εσωτερικό ε, ζήτημα διαχείρισης του ΕΛΚ. Και φυσικά υπάρχουν πολιτικές διαφορές, αλλά αν μια ομάδα γνωρίζει εκ των προτέρων ότι διαφωνεί με τον πυρήνα της έκθεσης, τότε προστεί οι διαπραγματεύσεις για τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Εφόσον καθόμαστε σε τράπεζα διαπραγματεύσεων για συμβαστικές τροπολογίες, φαντάζομαι ότι εννοείται ότι έχουμε μία ε, βούληση και διάθεση να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Αλλιώς ε, γιατί να το συζητάμε κιόλα. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ατυχές που δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση, αλλά εγώ προσπάθησα να συνεννοηθώ με όλες τις ομάδες και τώρα ορισμένοι με κατηγορούν να προσπάθησα να αποκλείσω οι αγνόησα μερικού. Ας χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που μας έμεινε για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα που θα είναι αποδεκτό από όλους, αλλιώς θα χρειαστεί να ψηφίσουμε, να λάβουμε θέση. Ακούσαμε, ακούσατε κυρία Άντιας Δεμέρα τις απαντήσεις της ηγήτριας. Θα σας παρακαλούσα να μην αρχίσουμε πάλι συζήτηση. Ευχαριστώ. Στη γλώσσα μου, στη γλώσσα του Θερβάντες, ο όρος με κονσουλτάρ, σημαίνει, η σημειολογική του έννοια τουλάχιστον είναι διευκολύνω τον αντίπαλό μου να εκφράσει τη γνώμη του. Καμία διαβούλευση δεν είχα μεταξύ μας, κυρία Βέλτ, δεν ζητήσα τη γνώμη μου ούτε του κυρίου Ντεγκράντες, καμία στιγμή. Αυτό που μου κάνατε δεν ήταν διαβούλευση, ενημέρωση μας κάνατε ότι τις τροπολογίες μας τις συνοψίζετε σε τρεις συμβαστικές τροπολογίες που δεν τις συζητήσατε με τους συντάκτες των αρχικών τροπολογιών. Μας επιβάλλετε ουσιαστικά τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν τις διαπραγματευθήκατε μαζί μας. Δεν είχαμε καμία διαβούλευση. Μην μας λέτε λοιπόν κύριε Εντβέλτ ότι μιλήσατε μαζί μου. Δεν μιλήσαμε για καμία από τις 38 μου τροπολογίες. Και είναι ψέμα να ισχυρίζετε κάτι τέτοιο. Δεν θέλω ως πρόεδρος της ε, Επιτροπής να πω ότι δεν έχει νόημα να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για τη διαδικασία. Υπάρχει δυνατότητα με την παράταση αυτή να καταλήξουμε σε ευρύτερη συμφωνία. Γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε την αναβολή της ψηφοφορίας για να δώσουμε περισσότερο χρόνο για τις διαβουλεύσεις και να καταλήξουμε σε μια πρόταση κοινή αποδοχής για το θέμα αυτό. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία της σας διάταξης. την ε, έκθεση του κυρίου Βος που αφορά τη συνολική προσέγγιση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείο 15. Τώρα αρχίζουμε να ψηφίζουμε επί της έκθεσης ΒΟΣ. Αρχίζουμε. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Διαδικαστικό. ότι Μπορούμε να ψηφίσουμε αν μπλοκ όλες τις προτάσεις συμβιβασμού, τις τροπολογίες συμβιβασμού. Oh, there more than that. Μπορείτε να το δεχτείτε. Να ψηφίσουμε μπλοκ τις περισσότερες τροπολογίες συμβασμού, τη μεγάλη πλειοψηφία τροπολογιών συμβασμού εκτός από 9, 34 και 36. 9, 34 και 36. Αυτό θέλουν και οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι αν δεν κάνω λάθος. Κύρκοπ. Και 20, και 20. Και 20. Οκ. Okay. Κάποιος άλλος. 18 και 20. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ψηφίζουμε λοιπόν. Unblock. Τους συμβιβασμούς όπως προαναφέρθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται όλες οι προτάσεις συμβασμού εκτός από τις προτάσεις που θα ψηφίσουμε τώρα. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση συμβιβασμού 20. 18 με συγχωρείτε, 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα. Τροπολογία 48. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογή 1 της Culture υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πολλές καταπίπτουν, πάρα πολλές καταπίπτουν. Μισό λεπτό. Σε ποια σελίδα είμαστε. 53. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για να δούμε, για να δούμε. 66, α, 56, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Ένα λεπτό. Δεν ξέρω ποιες καταπίπτουν και ποιες όχι. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε, ελέγξουμε καλύτερα. Τροπολογία 56. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 υπέρ 23 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Και περνάμε. Στο συμβασμό 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εξήντα τρία. Όχι με συγχωρείτε, 63 και 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 4 της Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 συμβασμού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ Α, με συγχωρείτε, ε, τροπολογία συμβασμού 8. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ. Έχει αποσυρθεί 82. 5 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε της Γιούρη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για να δούμε τώρα. Έξι της Γιούρη. Ξεχωριστή ψηφοφορία, πρώτη πρόταση, πρώτη ψήφος για την πρώτη πρόταση υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη πρόταση. Α, όχι. Καταπίπτει. Έξι ήτρε. Δεύτερη πρόταση. Υπέρ. Έξι της ήτρε. Δεύτερη πρόταση. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Well, 93. 93. Όχι, έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος, 91. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται μαζικά. 93. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7. Τη Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτηκε. 15 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 103. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. No, no. Amendment 8 της Ήτρε. Α, όχι, με συγχωρείτε, κάνω λάθος. Ο 8 της Επιτροπής Πολιτισμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι. Καλά. 9. Ήτρε. Θέλετε να ελέγξουμε την 8. Ελέγχουμε την 8 της Επιτροπής Πολιτισμού. Αρχίζει η ψηφοφορία. 8. Καλτ. Πέρας. Έχουμε έναν ε, επιπλέον από το ΕΛΚ. Έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ. Ποτέ, ποτέ δεν αρκούν. Maybe you are the one too many. Ίσως εσείς είσαστε υπεράριθμοι. Okay, then. Okay, we're taking off one vote for the EPP. Αφαιρούμε μία ψήφο από το ΕΛΚ. 22 έναντι 29. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην 9 της Ήτρε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Να σηκώνετε τα χέρια ευκρινώς διαφορετικά δεν βλέπουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε την καταμέτρηση. 17 ΙΜΚΟ αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 22-26. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 της Γιούρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 της Ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 της Ίμκο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 19 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 ήτρε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19 ΙΜΚΟ δεύτερη πρόταση. Μόνο τη δεύτερη πρόταση της 19 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12 της Επιτροπής Πολίτισμου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12 Ήτρε υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 12 ήτρε ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. ...24 έναντι 22 εγκρίνεται. Amendment 20 ΙΜΚΟ. 20 ΙΜΚΟ, το υπόλοιπο κείμενο υπόλοιπο κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 καλτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 ίμκο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 γιούρι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έχουμε μία ξεχωριστή ψηφοφορία. Όχι, όχι. We jump into 22 IMCO. 22 IMCO, πρώτο τμήμα. 22 IMCO. Σελίδα 16. Σελίδα 16. I think most of them have fallen. Νομίζω ότι έχουν καταπέσει οι περισσότερες. Fallen, fallen, fallen, fallen, up to all the way to amendment 20. Μέχρι την 22 της ΣΥΜΚΟ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται δεύτερο τμήμα, το δεύτερο τμήμα, νομίζω ότι απορρίπτεται. 136 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 κάλτ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 γιούρι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 ημκο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Ελέγχουμε την 146. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 28 έναντι 22. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ. 151 υπέρ. Ψηφίζουμε την ε, τροπολογία του Σταύρου. Εγκρίνεται. Και εσύ Σταύρο πρέπει να ψηφίσεις. 152 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβασμού 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 155. Όχι. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Προτρέχω 18 γιούρι. Πρώτη πρόταση. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19. Ήτρε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Γιούρι. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28. Προφορική. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Ήτρε. Υπέρ 21 Ήτρε, όχι της Γιούρη, της Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 Ήμκο. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 Ήτρε. Δεύτερη πρόταση υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 Ήμκο. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 της Ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Now, 33... 33 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 Ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 της Γιούρι Κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 26 της Γιούρι. Ελέγχουμε. Πέρας. 28 22 εγκρίνεται. 26 ήτρε τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 ΙΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 42 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τώρα πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τι θέλετε να ελέγξουμε? Την 42 της ΙΜΚΟ ελέγχουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία 42 ΙΜΚΟ ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται 35 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίθηκε, λυπάμαι, εγκρίθηκε. Ναι, είναι το θέμα της ανάτασης των χεριών. Πάντα το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οκτώ. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ένα. Ήμκο. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δώδεκα. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Ένα λεπτό. 27. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι αυτή τη φορά απορρίπτεται. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ. Απορρίπτεται. Μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος. 32. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά Κατά εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η μόνη που επιβιώνει είναι η έξι της ΣΥΜΚΟ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η τελευταία. Α, όχι, και η 44. Η εναπομείνασα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε στο κείμενο, το τεράστιο αυτό το κείμενο, όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Α, ηλεκτρονικά, με συγχωρείτε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Amounting to, let's see, 49 plus. 49, μία ψήφος κατά να συγχαρούμε τον κύριο Άξελ Βος. Και ταπεινά παρακαλούμε τον κύριο Βος να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Όχι πια τέτοια ψηφοφορία. Τέλος. Τώρα λοιπόν περνάμε. Έχουμε ακόμα μία ψηφοφορία. ως προς την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού ε, τα, τα συστήματα πληροφόρησης μεγάλης κλίμακας στο μία ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Κάρλος Κοέλιο. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Κοέλιο θέλει πάλι να, πάλι λάβει το λόγο πριν ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Καταρχήν για να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό με το Συμβούλιο και την Επιτροπή στην πρώτη ανάγνωση και όλες οι τροπολογίες σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα η οποία δεν επιτρέπεται ούτε η δημιουργία νέων συστημάτων χωρίς ε, νομοθετική διαδικασία, διορισμό μελών στα στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη Eurodac συμφωνήσαμε. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω να ψηφίσουμε αμπλόκ αυτόν τον συμβιβασμό έτσι ώστε αυτός ο οργανισμός να τεθεί σε λειτουργία του συντομότερο δυνατόν. Ψηφίζουμε λοιπόν. Αρχίζουμε. Κείμενο συμβιβασμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα όλες οι τροπολογίες καταπίπτουν. Ωραία, αυτό αντισταθμίζει την προηγούμενη ψηφοφορία. Ευτυχώς. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοέλιο. Τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. 43 υπέρ, 3 κατά. Να συγχαρούμε τον κύριο Κοέλιο για την εξαιρετική του εργασία. Και άλλο ένα σημείο έχουμε. Είναι μια έκθεση. Την έκθεση ως προς την αξιολόγηση για την οδηγία ε, για την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων. Μα ξεχάσαμε μία ψηφοφορία. Α, με συγχωρείτε, σημείο 17 δεν ψηφίσαμε, ναι δεν ψηφίσαμε την έκθεση φαγιών. Νόμιζα ότι είχαμε τελειώσει. Yes, I'm sorry, but I was, I was following my... Συγχωρείτε. Δεν υπήρχε αυτή η έκθεση στον κατάλογο ψηφοφοριών. Στο δικό μου κατάλογο έχουμε άλλη μια ψηφοφορία λοιπόν για, την... Για, τον... για την πρόταση απόφασης για έναν κατάλογο ταξιδιωτικών εγγράφων για τα εξωτερικά σύνορα εκεί όπου χρειάζεται θεώρηση και δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση κατά αυτού του καταλόγου. Τάνια Φαγιόν είναι η συγγήτρια και ψηφίζουμε το κείμενο. Ψηφίζουμε τη θέση της συγγήτριας υπέρ. Α, ηλεκτρονικά. Όχι, δεν χρειάζεται. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, Άρα εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο καθώς και την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Σαράντα υπέρ, κανένας κατά ομοφωνία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Φαγιόν. Λυπάμαι, ήμουν πολύ κουρασμένος και δεν είχα δει ότι έχουμε άλλη μια ψηφοφορία. Ωραία. Okay, okay. I've been reported. Okay, ενημερώθηκα. Ενημερώθηκα. Το τελευταίο σημείο της απογευματινής μας ημερήσιας διάταξη. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλώ, προσοχή. Το τελευταίο σημείο της απογευματινής μας ημερήσιας διάταξης είναι η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την έκθεση αξιολόγηση της οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων θα ακούσουμε την παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Διευθυντή κύριο Πρίβε. Αλλά κανονικά το σημείο αυτό έχει προγραμματιστεί για τις 6. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά μέχρι τις 6. Προτείνω μία ολιγόλεπτη διακοπή και σε ένα δεκάλεπτο επιστρέψτε στην αίθουσα για να συνεχίσουμε. We Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την κατανόησή σας. We thank you for your perseverance. Για την επιμονή σας, για την αντοχή σας, για την υπομονή σας, γιατί έχουμε και άλλο ένα θεματάκι. της Επιτροπής. Καλώς με τον κύριο Πρίβε, Διευθυντή της Γενικής ε, Διεύθυνσης Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μας παρουσιάσει την έκθεση Επιτροπής, έκθεση εξολόγηση οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Γενικό και μετά μπορεί να έχουμε και μερικές ερωτήσεις ε, λίγων λεπτών Έχετε το λόγο παρακαλώ κύριε Πρίβη. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και πάλι περιμένω με αγωνία και ανυπομονησία τις ερωτήσεις σας. Με χαρά να σας παρουσιάσουμε την έκθεση αξιολόγηση για την οδηγία περί διατήρησης δεδομένων. Όπως γνωρίζετε η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα μακρών διαβουλεύσεων, γραπτών, συνεισφορών, στατιστικών και ε, περίπτωση ολογίας ε, και ε, ακολούθησε και μακρά συζήτηση με τα κράτη-μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους εσκεμένα η έκθεση αυτή δεν είναι νομική ανάλυση. Δηλαδή δεν βγάζει συμπεράσματα για το αν και κατά πόσο η οδηγία με τη σημερινή της μορφή σέβεται ε, τις αρχές της, ε, ε, του αναγκαίου και του απαραίτητου και του αναλογικού. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας είναι απλή αξιολόγηση για το πώς λειτουργήσε στην πράξη η οδηγία, πώς εφαρμόζεται και αν χρειάζεται τροποποίηση. Η Επίτροπος Μάλστρομ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη διατήρηση δεδομένων ως ε, ένα εργαλείο για αποτελεσματική κοινή έρευνα στο συνολικό όφελος της δικαιοσύνης. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Επίτροπος είναι 100% ικανοποιημένη με το παρόν μέσον. Γιατί χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της διατήρησης δεδομένων. Θεωρούμε ότι υπάρχουν εξή τρεις λόγοι για να δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Πρώτον, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν ιστορικά ε, στην ποινική δίωξη και στην έρευνα. Αν δεν υπάρχουν κοινού κανόνες ε, δεν είναι σίγουρο ότι οι πάροχοι της υπηρεσίας θα μας τα διαθέτουν αυτά τα στοιχεία. Έχουμε δει κράτη-μέλη που δεν μετέφεραν ακόμα την οδηγία και έχουν σταματήσει ή εμποδίσει κοινέ διώξεις ε, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αυτή η νομοθεσία για τη διατήρηση δεδομένων γιατί τα κρατούσαν για πολύ μικρό διάστημα. Το δεύτερο, οι πάροχοι των υπηρεσιών ε, δικαίως περιμένουν ε, να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων δικαιοδοσιών στο εσωτερικό της εσωτερικής αγοράς και τρίτον οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε υψηλή ποιότητα προστασία και μόνιμη και διαρκή των προστατικών τους δεδομένων και προστασία του δικαιώματος ε, της ιδιωτικής τους σφαίρας όπου και να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βεβαιωθούμε ότι και αυτά τα και τα τρία ε, ως στόχοι πληρούνται. Γιατί χρειάζεται και αν χρειάζεται μεταρρύθμιση τη οδηγίας. Τα περισσότερα κράτη-μέλη εκφράζουν την ικανοποίησή τους στη διαδικασία διαβούλευση με την παρούσα οδηγία γιατί ε, ε, επιτρέπει πολλή ευελιξία για τον τρόπο με τον οποίο ε, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να διαβιβάζονται και να χρησιμοποιούνται. Αλλά πολλά κράτη επίσης έχουν γνωρίσει δυσκολίες στη μεταφορά της οδηγίας και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σε τρεις περιπτώσεις, Ρουμανία, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία, τα συνταγματικά δικαστήρια έχουν απορρίψει τη μεταφορά στην ένωμη τάξη ε, της χώρας. Αντίστοιχα συμβαίνουν στη Βουλγαρία και την Κύπρο και σε μια έκτη χώρα, στην Ουγγαρία, που εκκρεμεί ακόμα η υπόθεση στο συνταγματικό δικαστήριο. Ε, στο μεταξύ, μάλλον τελικά το ΔΕΚ θα κληθεί να αποφανθεί για το νόμιμο ε, της ε, οδηγίας ε, όταν εκδικαστεί υπόθεση για την οποία προσέφηκε μια ομάδα δικαιωμάτων του πολίτη από την Ιρλανδία σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα της αναλογικότητας αφήνει ένα περιθώριο χειρισμό στα κράτη-μέλη για τον τρόπο ε, που θα εφαρμόζουν ε, αυτή τη δυνατότητα ε, Ποιο θα έχει πρόσβαση, ποιο θα φυλάσει τα δεδομένα, αν θα έχει πρόσβαση η δικαιοσύνη, η αστυνομία, άλλε διοκτικέ αρχές. Ε, θα πρέπει να βλέπουμε πώς αλλάζουν οι αξιόπινες περιφορές και οι τεχνολογίες, πώς έχουν αλλάξει τις επικοινωνίες τα τελευταία πέντε χρόνια και να προβλέπουμε για την επόμενη πενταετία με δεκαετία ορισμένα κράτη-μέλη επί ζήτησαν μια ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση για ανώνυμες κάρτες κινητής τηλεφωνίας SIM. Ε, το θέμα των smartphones και του διαδικτύου επίσης ε, θα χρειαστεί απαντήσεις και θα πρέπει να αναρτηθούμε κατά πόσο το παρόν σύστημα διατήρησης δεδομένων συνεχίζει να είναι επίκαιρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση του φυσταμένου πλαισίου. Αρχίσαμε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους για να τους συζητήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και στις 8 Ιουνίου. Και αντίστοιχα εργαστήρια θα γίνουν με ε, τους ενεχομένους, με τις διοκτικές αρχές, με τους κλάδους, με τη δικαιοσύνη, με τα κρατημέλη της ερχόμενες εβδομάδες έχουν προγραμματιστεί αυτές οι συζητήσεις. Ποιες είναι δεχόμενες τώρα επιλογές και δυνατότητες που έχουμε μεταρρύθμισης. Θεωρητικά, ας πούμε, Μία επιλογή θα ήταν το status quo, να διατηρηθεί ως έχει η κατάσταση, αλλά να συνεχίζεται ε, η δράση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προσφεύγει επί παραβάση. Όπως σας είπα, κάποια κράτη-μέλη ζητούν να παραμείνει η κατάσταση ως έχει και πολλά μάλιστα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα προστασίας δεδομένων, ιδιωτική ζωής και κάποιες αλλαγές και σημερινές και επόμενες δεν μπορεί να διατηρηθεί το καθεστώς ως έχει. Το δεύτερο είναι να ακυρωθεί συνολικά, να καταργηθεί οδηγία και να επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να ε, επιλέγουν τη δική τους προσέγγιση. Αυτό επιτρέπεται από την οδηγία ε, για την ιδιωτική ζωή στο άρθρο 15. Και η τρίτη εναλλακτική λύση που θα προτιμούσαμε εμείς είναι να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε καλύτερα στάνταρ αναλογικότητας χωρίς να διακυβεύεται η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του μέσου. Δεν τίθεται θέμα εναρμόνισης ε, για την εναρμόνιση. Δεν είναι αυτός σκοπός. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις στον κλάδο και στα θεμελιώδη δικαιώματα της οδηγίας ε, ε, ανταποκρινόμενη στο στόχο της. Γι' αυτό τα συζητούμε με τα κράτη-μέλη, τα υπέρ και τα κατά, τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογή ε, των περιόδων διατήρησης δεδομένων και των ασφαλιστικών δικλείδων. Αλλά δεν διστάζουμε ε, να ζητήσουμε και άλλες προτάσεις για τη διατήρηση των δεδομένων. Επιτρέψτε μου σύντομα να αναφερθώ σε κάτι ακόμα. Μέχρι να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, τι θα κάνουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το ισχύον πλαίσιο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να βεβαιωθούμε ότι η παρούσα οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων μεταφέρεται σωστά στην ένωμη τάξη τη κάθε χώρα. Επειδή έχουμε παράπονα και καταγγελίε για το κατά πόσο είναι απαραίτητη μια τέτοια οδηγία θα πρέπει να συνεχίζουν να δίνουν στατιστικά στοιχεία βάσει του άρθρου 10, αλλά και ποιοτικά ε, στοιχεία και πιστήρια και τεκμήρια για να δούμε τελικά στην πράξη ποιο ήταν το απτό χειροπιαστό αποτέλεσμα και τι σημαίνει η διατήρηση δεδομένων και ποια ήταν αυτά που ε, βοήθησαν, ε, που ήταν κρίσιμα για να εξεχνιαστεί ένα έγκλημα και να προστατευτεί ή να αθωωθεί ένας αθώος τελικά. Επίσης, Πρέπει να δούμε τι ισχύει και με τους ε, παρόχους των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει όλα αυτά τα θέματα και θα κάνει τις προτάσεις της. Ε, κατά τη διάρκεια του θέρους θα κάνουμε μια μελέτη σκοπιμότητας βάσει αυτών που σας ανέφερα προς τις επιλογές. Θα επιλέξουμε μια δυνατότητα για τη μεταρρύθμιση και θα ζητήσουμε και μία μελέτη για την, εκτίμηση, την αίσθηση που έχει το κοινό για τα θέματα αυτά και ποια μοντέλα υπάρχουν για τη διατήρηση δεδομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να ολοκληρώσω, για να είμαι πλήρη στην τοποθέτησή μου, κύριε Πρόεδρε, για τα κράτη-μέλη Κίνα που μέχρι τώρα δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία, είναι πολύ λίγα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφύγει στο δικαστήριο επί παραβίαση, επί παραλήψη. Ευχαριστώ. Άρχεται η συζήτηση, παρακαλώ. Ποιος θέλει το λόγο. Κύριε Έντβελτ. καλύτερα να δώσετε πρώτο λόγο στον κύριο Άλβαρο που ήταν ο προηγούμενος συγητής. Θα είμαι λακωνικότατη γιατί είχαμε εκτενέστατη συζήτηση για το ίδιο θέμα την περασμένη εβδομάδα στο σεμινάριο και μερικοί εξεπλάγησαν ότι γιατί παρά τις πολυάριθμες κριτικές για την οδηγία αυτή διατήρηση δεδομένων, ακόμη και από το EDPS, επαναλαμβάνει σαν σπασμένο γραμμόφορο να επαναλαμβάνει πόσο καταπληκτική είναι αυτή η οδηγία, αντί να ακούσει τις επικρίσεις και να προβληματιστεί και αυτή για το κατά πόσο είναι απαραίτητη με τέτοια οδηγία. Γιατί αν συγκεντρωθούν τα στοιχεία για τον παραμικρό για τον κάθε πολίτη ε, μπορεί να, είναι να γίνει ασφαλέστερη κατάσταση, αλλά δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Και με εντυπωσιάζει που δεν ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις επικρίσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την τελευταία διετία δεν άκουσα ούτε έναν πιστικό και ευνόητο λόγο για τον οποίο δικαιολογείται αυτή η οδηγία. Δεν ξέρω πώς απαντά στις επικρίσεις του EDPS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν μιλάμε για μομφές ακτιβιστών εδώ. Μιλάμε για ένα γραφείο που προβαίνει σε πολύ αμερόληπτη και αντικειμενική και τεκμηριωμένη ανάλυση της οδηγίας. Πώς ε, καταρρύπτεται αυτές τις επικρίσεις. Κύριε Σάλβαρ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ε, διαφωνούμε σε αυτό το θέμα, είναι κοινό μυστικό. Καλό θα ήταν όμως να κάνουμε μια συζήτηση αντικειμενική για την οδηγία αυτή. θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί και μάλιστα οπωσδήποτε και όχι να είναι η κασία αυτό και η υπόθεση. Ε, θέλω να ρωτήσω το εξή που με ενδιαφέρει. Έχουμε κάποια εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αμοιβαία είναι και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διοκτικές αρχές πάντα μας εξηγούν πόσο απαραίτητη είναι η διατήρηση δεδομένων. Μπορεί να μας αναφέρει μία περίπτωση, εκτός από την περίπτωση της ε, Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της παιδικής προνογραφίας. μία διασυνοριακή περίπτωση όπου να είχαν πραγματικά αποτέλεσμα, ε, να ήταν ε, αποδεδειγμένα απαραίτητη η ακράτηση, αυτή η διατήρηση. Γιατί η γερμανική αστυνομία δεν μας ε, δίνει στοιχεία. Ε, ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της διατήρησης δεδομένων διασυνοριακή συνεργασία. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο. Αυτό το καιρό έχει προσφύγει η Ιρλανδία στο προδοδικείο ε, για το θέμα του πόσο συνάδει αυτό με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το χάρτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συναντήσει άτυπα το πρωτοδικείο γιατί θα ήταν πραγματικά έτσι κάπως πρόβλημα και θα μας εξέθετε ε, εάν ε, αποφαινόταν το πρωτοδικείο όπως ε, το Ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο και έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν συνάδει με το, το χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων στην Ένωση. Έτσι θα ήταν κάπως εκτεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω τη λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να προχωρήσει την προσφυγή κατά των κρατών γνωρίζοντα ότι θα αναθεωρηθεί η οδηγία. Μιλώ για τη Γερμανία ανεξάρτητα από ε, το καθεστώς των Υπουργείων ε, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Επροκειμένων Ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο καιρό χρειάζεται η νομοπαρασκευή σε ένα κράτο μέλο και να περάσει από την Bundestag και μέχρι ε, να γίνει αυτό θα έχει αναθεωρηθεί η οδηγία και θα ζητείτε νέος νόμος. Πέρα από το θέμα της γραφειοκρατίας, το θεωρείτε τόσο πολύ απαραίτητο να συνεχίσετε τη διαδικασία προσφυγής επί παραλήψη. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί καθυστέρησα, δεν άκουσα τις ε, εναλλακτικέ που προτείνατε. Το quick freeze και το data preservation ε, σκέφτεστε να το συνδυάσετε. Υπάρχει και μια τέτοια πιθανότητα ή δυνατότητα στην αθεώρηση. Και ένα τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν πρόθυμη να έρθει σε μια συζήτηση στην Ολομέλεια. Γιατί είναι άλλες οι ευαισθησίες σήμερα στο Κοινοβούλιο από το 2005. Θα εξακολουθήσει να αρνείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Γιατί καλό θα ήταν πριν την αναθεώρηση να γίνει ε, σε κανονικά συζήτηση στην Ολομέλεια. Δεν ξέρω να το θέσει και υπόψη τη διάσκεψη των Προέδρων ο προεδρό μας. Και τελειώνω επειδή μακρηγόρησε. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζει η Ελλάδα τη διατήρηση των δεδομένων. ότι τα στοιχεία που συλλέγονται στην Ελλάδα μπορούν να διατηρούνται μόνο στην Ελλάδα. Αυτό συνάδει με το πνεύμα και το γράμμα της οδηγίας ή θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ότι ε, παραβιάζεται η ευρωπαικη επιτροπη οτι ε κυκλοφορία των δεδομένων. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Άλβαρο, το σημείωσα, αλλά θα προτιμούσα να μου στέλνετε και mail με την διατύπωση που προτείνατε, ώστε να τη διαβιβάσουμε στην ε, διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών. Ο κύριος Βός. Μία ερώτηση προς την ίδια κατεύθυνση με εκείνη του Αλεξάνδρου Άλβαρο. Έχει νόημα πραγματικά να συνεχίσετε ε, την προσφυγή στο δικαστήριο και να αναγκάσετε τη Γερμανία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να περάσει νόμο, ενώ προβλέπετε να θεώρηση οδηγίε που θα χρειαστεί νέο νόμο. Και ένα ακόμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να, το απαντήσετε εσείς. Αυτά τα τρία συνταγματικά δικαστήρια έχουν την ίδια αιτιολογική ε, σκέψη, ας πούμε, δικαιολόγηση απόφασης και ως προς τη διάρκεια. Έχουμε εμπειρία από το παρελθόν για το πόσο καιρό θα πρέπει να κρατούμε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή κάπου ακούμε ότι αν μετά από τρεις μήνες ε, δεν βοήθησε σε κάποια δίωξη, δεν έχει νόημα μετά την παρέλευση του τριμήνου. Έχετε όμως εσείς εμπειρία, έτσι, ποιο χρονικό διάστημα κρίνεται μου. Αν δεν τα ξέρετε εσείς αυτό, να ρωτήσουμε αλλού. Έχετε το λόγο κύριε Κύρκο. Ευχαριστώ. Έχω δύο σχόλια. Το ένα αφορά τις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. και τι ακριβώς λέμε, αν συμφωνούμε στην ορολογία, γιατί χρησιμοποιούμε με την ίδια γλώσσα τα αγγλικά, αλλά ως προς τα νοήματα ίσως ε, υιοθετούμε διαφορετική ερμηνεία. Για παράδειγμα, προστασία των ε, συμφερόντων, ασφάλεια των πληροφοριών. Έχουμε κάποιες βασικές έννοιες εδώ. Είναι σίγουρο ότι τις αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο και τις κατανοούμε με τον ίδιο τρόπο, γιατί και εμείς είχαμε προβλήματα ε, και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει, υπάρχουν παρεξηγήσεις μερικές φορές μεταξύ ημών και των Αμερικανών για ορισμένα από αυτά τα θέματα. Είναι προχωρημένη η σύγκριση στις θέσεις, στις προσεγγίσεις που υιοθετούμε η ΜΕΝ και η ΔΕ και ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς αντιλαμβάνονται εκείνες αυτές τις έννοιες. Μιλούμε για φύλαξη δεδομένων ή διατήρηση δεδομένων ή πληροφοριών. Μερικοί μίλησαν για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τέτοια διατήρηση. Δεν είναι το μόνο κριτήριο όμως που ενδιαφέρει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει όχι μόνο η διάρκεια της διατήρησης, αλλά και πώς ε, φυλάσσονται αυτές ε, οι πληροφορίες, πόσο ασφαλές είναι το σύστημα που τις ε, διατηρεί, τι εχέγγυα δίνονται, τι ασφαλιστικές δικλείδες και τι χρήση επιτρέπεται στις πληροφορίες αυτές και ποια η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Αυτό είναι εξίσου σημαντικά με, την, με τη διάρκεια της διατηρήσης, το χρονικό διάστημα, για να μην πω και πιο σημαντικά. Πιστεύετε ότι οι υφιστάμενες προτάσεις επαρκούν για να προστατεύσουν και από αυτή τη σκοπιά τους πολίτες. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η αξιολόγηση είναι κάτι που διάβασα με μεγάλη προσοχή όπως και άλλα έγγραφα και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι πήγαν μερικά πράγματα στραβά σε αυτή τη διατήρηση δεδομένων. Και ίσως ένα από τα λάθη που κάναμε ήταν ε, τόσο ταχεία ε, διαδικασία για τη νομοθεσία. Αν δούμε πόσα χρήματα ε, χρειάστηκαν και μόνο από την πρακτική διάσταση από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύων από ε, τηλεφωνικές εταιρείες επικοινωνίας για να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία τουλάχιστον στη Γερμανία νομίζω ότι οι επενδύσεις είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη ε, εφαρμογή ε, αυτής της νομοθεσίας. Αν δείτε λοιπόν πόσα χρήματα έχουν εκταμιευθεί εκεί, είναι μεγάλο μυστήριο η όλη υπόθεση. Και τη βλέπουμε σχετικά σαφώς ε, ότι με τον τρόπο που έχουν αποφασιστεί αυτά τα πράγματα δεν έχουν νόημα, δεν βοηθούν ουσιαστικά στην ποινική δίωξη και γενικότερα κινούνται σε έναν εφέλωμα και σε μια θολή κατάσταση ε, για τον τρόπο που εφαρμόζονται. Είναι τελείως ε, αλλοπρόσαλη ε, και πάρα πολύ διαφορετική η εφαρμογή στα κράτη-μέλη που το έχουν εφαρμόσει αυτό και έχουν μεταφέρει την οδηγία και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ε, καθόλου σαφής γνώμονας για την αναλογικότητα και για τη σκοπιμότητα καν αυτής της νομοθεσίας. Και σε ό,τι αφορά τις νομικές προϋποθέσεις και το πλαίσιο, ακούσαμε ότι υπήρξαν συνταγματικά δικαστήρια σε ορισμένα κράτη-μέλη που απέρριψαν αυτή τη νομοθεσία, είτε τον εφαρμοστικό νόμο, είτε την οδηγία και την ίδια. Τι θεώρησαν ε, αντισυνταγματική στις χώρες τους. Και βασίστηκαν στα στοιχεία που έχουμε, τα συντάγματα των κρατών μελών, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ΕΣΔΑ και την ομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα γνωρίζαμε από το παρελθόν και τα αναφέραμε ξανά και ξανά. Και επιτέλους έχει έρθει η ώρα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ομολογία αυτή να την πάρει υπόψη της και τα μέτρα που λαμβάνει να τα προσανατολίζει σε αυτό το πλαίσιο και να διατηρείται εντός αυτού του πλαισίου. Είναι νομίζω καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό. Να φροντίσει αυτό το πλαίσιο να είναι συνεκτικό στην Ένωση, το νομικό πάντα. Διότι οι πολίτες στην Ευρώπη, αλλά και οι πελάτες στην Ευρώπη, ε, των παρόχων επικοινωνιών δεν μπορούν να περιμένουν χρόνια ολόκληρα μέχρι να το λύσει αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να έχουν ασφάλεια δικαίου και να μπορούν να λειτουργήσουν και να ε, δικαιωθούν. Αυτά είναι απαράδεκτα κατά την άποψή μου και ρωτώ. Πότε σκέφτεστε να φέρετε πρόταση για την αναθεώρηση και θα συνεργαστούμε ενεργά. Ευχαριστώ κύριε Κορατσαμπίλτ. Ευχαριστώ. Με εξέπληξε η ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι εξετάζει ακόμη και τη διατήρηση της ε, μέχρι τώρα κατάστασης. Νομίζω ότι είναι αντιφατική αυτή η συμπεριφορά γιατί ε, μερικές χώρες δεν έχουν ε, μεταφέρει ακόμη την οδηγία αυτή στην εσωτερική τους αναμετάξη μετά από ψηφοφορία στα κοινοβουλιά τους και πολλές φορές και από την κοινή και από τα δικαστήρια και από τα εθνικά κοινοβούλια ε, προκύπτουν ε, βάσιμες επικρίσεις για θέματα ιδιωτικής ε, ζωής, για δυσανάλογη χρήση του συστήματος αυτού, για υπερβολική παρεμβατικότητα, για έξι, από δύο έξι χρόνια διακύμαση του χρόνου διατήρησης, άλλες χώρες είναι υπέρ της επιμήκης, άλλες όχι, για πόσο σοβαρά εγκλήματα θα πρέπει να επιτρέπεται ε, τέτοια διατήρηση. Όλα αυτά τα σημεία δείχνουν ότι το ζήτημα επήγει και θα πρέπει να διαθετηθεί. Περιμένουμε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς προτίθεται να θεωρήσει την παρούσα οδηγία προκειμένου να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ε, ανησυχίες και τον προβληματισμό. Γιατί φαίνεται ασυνεπές να συνεχίζετε την ε, τυπική διαδικασία ασκήσεων προσφυγών επί παραβάση κατά χωρών που δεν την έχουν μεταθέσει αυτήν την οδηγία, αλλά κοφεύεται στις ε, ε, εύλογες ανησυχίες και δημοκρατικά εκλεγμένων σωμάτων και των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών. Η κυρία Λάτφορτ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη σύγχυση και πριν από έξι χρόνια παρόμοια κατάσταση είχαμε. Σαν να μην έχουμε προχωρήσει καθόλου. Και δεν το λέω προσωπικά αυτό προς τον κύριο Πρίβε. Υποτίθεται ότι η οδηγία προτείνει απεριόριστη νομική ασφάλεια και προβλεψιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει τη δυνατότητα διατήρησης δεδομένων σε διάφορες χώρες μέλη. Περιορισμένη λοιπόν, συγγνώμη, αυτή η προστασία, η νομική ασφάλεια, όπως ακούσαμε αλλά υπάρχει διακριτική ευχαίρεια για την υιοθέτηση των μέτρων αυτό με βάση το άρθρο 51 και το θέμα ε, ακριβώς εξαιτία τη διακριτική ευχαίρειας καθιστά την αξιολόγηση για την εφαρμογή της οδηγία αυτής και το κατά πόσο εφαρμόζεται μάλλον δύσκολη. Άρα με τι δικαίωμα προσφεύγεται αφού είναι αμφίβολη η αξιολόγηση τη σωστή εφαρμογή είναι σαν να μιλάμε με ακαδημαϊκά παραδείγματα, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Είχαμε παρόμοια α, περίπτωση στο παρελθόν με μια νομοθετική πράξη και είπαμε να αποφευθεί η επανάληψη που είχαμε την, την νομοθετική πράξη για τα επικίνδυνα σκυλιά. Ε, συμμετείχατε και εσείς στην εκπόνηση. Α, συγγνώμη, το είχα ξεχάσει. Συγγνώμη που το ανέφερα. Δεν είχα δεν θυμόμαι τη δική σας εμπλοκή στο θέμα αυτό. Πάντως αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ε, νομοθετικής, ε, άστοχης νομοθετικής δράσης. Φαντάζομαι ότι το κάνετε υπό πίεση των πρεσταμένων σας. Φαίνεται ότι η οδηγία αυτή είναι η ευρωπαϊκή εκδοχή της, ε, του νόμου για τα επικίνδυνα σκυλιά. Τελικά αναφέρθηκε ως βεβαιασμένη ε, νομοθεσία ως αντίδραση της ε, τότε κυβέρνησης στην, ε, στις βομβιστικές επιθέσεις του Λονδίνου του Ιουλίου. Πραγματικά ήταν εσπευσμένη διαδικασία, βεβαιασμένη, δεν έγινε ο απαραίτητος έλεγχος και τελικά ήταν τελείως αποτυχημένη η εφαρμογή του νόμου αυτού για τα επικίνδυνα σκυλιά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι τέτοιο θυμίζει η ισχύουσα οδηγία. Αν το ΔΕΚ ήταν έντιμο θα έπρεπε να αναστείλει το άρθρο 95 γιατί ε, περί αυτού πρόκειται. Αυτό κάνει η οδηγία ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση δεδομένων για επικίνδυνα εγκλήματα. Τελικά η οδηγία δεν προβλέπει ούτε την πρόσβαση δεδομένων, ούτε τη χρήση των δεδομένων, ούτε την ανταλλαγή των δεδομένων. Και εξού και η έλλειψη νομικής σαφήνειας και ασφάλειας για τους ε, χρήστες. Πραγματικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό, δεν μας έβαλε αυτή στο, στο μπέρδεμα, αλλά περιμένουμε τη βοήθειά της για να ξεφύγουμε από αυτό το μπλέξιμο. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρετε. Θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ΔΕΚ για την Ιρλανδία, αλλά σίγουρα κάτι θα πρέπει να γίνει. Τουλάχιστον ως προς αυτό να συμφωνήσουμε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει για να ξεφύγουμε από την κατάσταση που, στην οποία βρισκόμαστε τώρα από μια πιο ιδανική περίπτωση. Γιατί πραγματικά εμείς είναι που πληρώνουμε τα σπασμένα, γιατί εμείς είμαστε οι πελάτες, οι χρήστες τελικά αυτού του συστήματος. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πρίμπε για να απαντήσει στις ερωτήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, φοβάμαι ιδιαίτερα τα σκυλιά. Θα πρέπει να σας ε, το ομολογήσω αυτό και θα θεωρούσα ε, το νόμο πολύ κακό αν αφορά μόνο τα μεγάλα σκυλιά, γιατί εγώ φοβάμαι ακόμα και τα μικρά. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω να αποφύγουμε παρόμοια λάθη ως προς το νόμο για την διατήρηση δεδομένων. Έχουμε μόνο πέντε λεπτά, γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα σύντομος και να δώσω απαντήσεις σε όλους. Μετά από αυτή την μακρά προετοιμασία αυτής της έκθεσης, η Επιτροπή έφτασε στο συμπέρασμα και μπορεί να διαφωνήσετε βεβαίως ότι πολλά επιχειρήματα προβλήθηκαν ως προς το ότι είναι ένα πολύ σκόπιμο και εύλογο μέσο. Ε, ποτέ δεν βρίσκεται ε, ρηξικέλευτα σχόλια ή σχόλια ας πούμε ακραία, θετικά ακραία του τύπου «αυτό είναι εξαιρετικό», ε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί μια ουσιαστική αλλαγή και ούτω καθεξής. Στο Συμβούλιο είχαμε την εντύπωση ότι θα είχαμε μια ε, ειδική πλειοψηφία κατά αυτής της οδηγίας, γιατί υπάρχει μεγάλη διχογνωμία σε επίπεδο κρατών μελών. Θεωρήσαμε ότι η έκθεση έλαβε υπόψη όλες τις πτυχές αυτού του δυσχερούς ζητήματος και δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν λάβαμε υπόψη και τα σχόλια του επόπτη κατά το σεμινάριο του Δεκεμβρίου. Θα σας μιλήσω για περιπτώσεις. Πολλές φορές μου λέτε ότι αναφέρομαι σε πολλές αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να το ελέγξω. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ε, είναι χρήσιμο αυτό το μέσο όταν έχουμε να κάνουμε με διασυνοριακές περιπτώσεις για την προστασία των δεδομένων, ακόμα και αν αυτό το μέσον καλύπτει τα κράτη-μέλη αποκλειστικά. Θα πρέπει όμως να το ελέγξω. Τώρα ως προς τις ε, διαβουλεύσεις με δικαστήρια ενδεχομένως. Αυτό θα το σύστηνα. Δεν θεωρώ ε, ένα δικαστήριο, σοβαρό, σοβαρό δικαστήριο αν δεχτεί ένα τέτοιο αίτημα. Ως προς τις εκκρεμείς διαδικασίες ε, παράβασης, Εάν κάτι πρέπει να βελτιωθεί στην τρέχουσα νομοθετική διαδικασία, αυτό σημαίνει ότι το θέμα αυτό πρέπει να φτάσει στο νομοθέτη το ταχύτερο δυνατό. Όμως δεν θέλουμε να εκτεθούμε σε επικρίσεις ότι κινηθήκαμε με ιδιαίτερη σπουδή. Γι' αυτό θα γίνουν οι διαβουλεύσεις καθώς και μελέτη αντικτύπου για να δούμε κατά πόσο πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Θα χρειαστεί λοιπόν λίγος χρόνος. Από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ε, θεωρήσει ότι πρέπει να σταματήσει τις διαδικασίες ε, επί ή κατά παράβαση σε σχέση με ορισμένα κράτη-μέλη τη στιγμή που έχει καταβληθεί προσπάθεια μεταφοράς της οδηγίας εδώ και αρκετά χρόνια. Από την άλλη πλευρά, αν λάβετε υπόψη την τρέχουσα οδηγία και την ε, τελευταία σελίδα αυτής της αξιολόγησης όπου βλέπετε προς τα πού κινούνται τα πράγματα, τότε βλέπετε ότι μπορεί να μεταφερθεί η τρέχουσα οδηγία έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μην χρειαστεί να επανανομοθετήσουν εάν αλλάξει η οδηγία στο μέλλον. Δεν αποκλείεται βεβαίως κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και αναγκαίο για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, μετατάξει την οδηγία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ε, Γερμανίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέφερε στην απόφαση του ότι ναι, υπήρξαν επικρίσεις, αλλά υπάρχουν δυνατότητες μεταφοράς ε, αυτής της οδηγίας, έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με το εσωτερικό δίκαιο. Είδαμε με μεγάλη προσοχή τις αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν θέματα εσωτερικής τάξης Και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να επεκταθούμε περαιτέρω σε αυτό το ζήτημα. Ε, λάβαμε υπόψη την απόφαση των συνταγματικών δικαστηρίων σε σχέση με θέματα εσωτερικής νομοθεσίας. Ως προς τη νομική βάση, κατανοώ τις επιφυλάξεις σας, είναι και το μόνο θέμα το οποίο διευκρίνησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου σε σχέση με το άρθρο 95 ως νομική βάση, όπως όρισε το ΔΕΚ. Νομίζω πρέπει να σταματήσω ναι. εδώ γιατί ναι. βιάζεστε. Τώρα πότε θα υποβάλει πρόταση η Επιτροπή δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εργαζόμαστε εντατικά ε, με διαβουλεύσεις και μία μελέτη επιπτώσεων θα χρειαστεί οπωσδήποτε, η οποία είναι υπόθεση μηνών, υποθέτω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρίπε. Αυτά Αυτά επί του παρόντος νομίζω ότι η εισήγηση αυτή για την κατάσταση, την υφιστάμενη κατάσταση είναι επαρκής και θα διακόψουμε τη συνεδρίασή μας μέχρι αύριο στις 9. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο στις 9. Γεια σας.